Well, thank you very much. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας με μεγάλη χαρά. Χαιρετίζω τον ε, ε, Γενικό Γραμματέα της Ελβετίας για τα εξωτερικά θέματα, τον κύριο Ρωσιέ, που θα αντιμετωπίσει θέματα τα οποία ξεπερνούν βέβαια το στενό πλαίσιο των διμερών σχέσεων που ακούσαμε χθες. και θα σταθεί σε ορισμένα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία και θα εξετάσει πώς μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο στα θέματα αυτά και τούτου λεχθέντος θα ήθελα να προσκαλεί να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το προνόμιο και την τιμή που μου κάνετε να σας παρουσιάσω τους κεντρικούς άξονες της εξωτερικής μας πολιτικής. Όπως κάθε χώρα η Ελβετία έχει τις δικές της αξίες και αρχές οι οποίες συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών της και των εθνών που την συναποτελούν. Αυτά είναι εγγεγραμμένα στο Σύνταγμά μα, είναι οι αρχέ τη αλληλεγγύη, τη καταπολέμηση τη φτώχεια, ε, του σεβασμού τη δημοκρατία, τη ειρηνική συνύπαρξη και τη ε, συντηρήση των φυσικών πόρων. Επιτρέψτε μου να περάσω από το ειδικό στο διεθνέ και στο πιο ε, γεωγραφικά εντοπισμένο. Ξέρετε ότι η Ελβετία έχει πολλού φυσικού πόρου, αλλά είναι στραμμένη και προ το εξωτερικό. Χρειαζόμαστε απελευθέρωση των συναλλαγών απελευθέρωση ε, που μέσα από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης μπορεί να προκαλέσει απώλειες ή ωφέλη για τους μεν και τους δε. Η ουσία λοιπόν είναι να μειώσουμε τα αρνητικά στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Υπό αυτή την έννοια η Ελβετική Βουλή αποφάσισε να φτάσει στο 0,5% την ε, κρατική βοήθεια προς ανάπτυξη η οποία έχει δύο, ε, ένα διτό προσανατολισμό. Πρώτα απ' όλα εντοπίζεται στα ευάλωτα περιβάλλοντα ξέρουμε. Ε, περίπου η μισή από την συνολική μας βοήθεια για τα ερχόμενα χρόνια από το 1 τρίτο που ήταν πριν και βεβαίως την ε, αναπτυξιακή βοήθεια μαζί με αρχές διακυβέρνησης πλέον, δηλαδή την δημιουργία θεσμικού κράτους σε ευάλωτα περιβάλλοντα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Μαλί, όπου ε, δραστηριοποιήθηκε η Ελβετία στα πλαίσια της ανθρωπιστικής κρίσης που υπήρξε εκεί με προσπάθειες για την ανάκαμψη της χώρας, τη στήριξη υποστήριξη τη διακυβέρνηση των φορέων τοπική αυτοδιοίκηση στον βορρά τη χώρα, γιατί ξέρετε ότι στον βορρά τη ε, χώρα αυτή είναι ε, εντοπισμένα τα αίτια που ε, πλήττουν τη σταθερότητα τη χώρα και τη γενικότερη περιοχή του Σαχέλ. Η Ελβετία λοιπόν εντοπίζεται στο βορρά του Μαλή και προσπαθεί με ρόλο διαιτησία και διαμεσολάβηση να στηρίξει όσα ε, ε, κάνουν τα κράτη της Δυτικής Αφρικής ως κοινότητα για την σταθεροποίηση του Ουακαντουγκού. Ε, κατά τα άλλα, η Ελβετία συμμετέχει στις διαβουλεύσεις του ΟΗΕ για την ε, υλοποίηση των προτεραιοτήτων για την, ε, με την ατζέντα του 2015. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του νερού, διότι η, Ελβετία δεν έχει πολλούς μεν φυσικούς πόρους, αλλά έχει πάνω απ' όλα νερό. Αυτό ε, είναι ένα από τα πιο πλούσια στοιχεία που διαθέτουμε, πολλούς υδάτινους πόρους στην επικράτειά μας. Έτσι λοιπόν στην περιοχή των συνόρων έχουμε ιδιαίτερου μηχανισμούς για την ε, διαχείριση των φυσικών πόρων πέρα του νερού και ε, με συστήματα διαβούλευσης δύο ε, παραδείγματα η κοιλάδα του Φραγκανάτ στο Ουσμπεκιστάν και μια και επίσης μια ακόμη κοιλάδα μεταξύ της Συρίας και του Λιβάνου, ένα σημείο που και αυτό αποτελεί προτεραιότητα για μας. Η προσέγγιση μας όμως ε, καταρτίζεται και σε διμερές επίπεδο με το αποτύπωμα που έχουμε δημιουργήσει στο Βιετνάμ, όπου έχουμε υποχρεώσει χιλιάδες ε, ε, παραγωγούς καφέ να μειώσουν κατά 70% το, την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιούν. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δεσμεύεται η Ελβετία στους διεθνείς της στόχους. Βεβαίως η παγκοσμιοποίηση σημαίνει και κανόνες δικαίου. Γι' αυτό η Ελβετία όπως ξέρετε στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και του ανθρωπιστικού δικαίου έχει ιδιαίτερη δράση μαζί με την ε, σύμβαση της Γενέβης. Νομίζω δύο άξονες εδώ πρέπει να εντοπιστούν. Πρώτα απ' όλα η ανάγκη να έχουμε καλύτερη υλοποίηση του ανθρωπιστικού διεθνούς δικαίου βάσει της γενικής συνένεσης που υπάρχει και των ε, γενικών αρχών του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι τώρα η υλοποίηση είναι πλημελής. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί ε, ο σεβασμός του ανθρωπιστικού δικαίου ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ένα σύστημα συμμόρφωσης, ένα σύστημα ελέγχου και με εθνικές εκθέσεις. Ένα παράδειγμα υλοποίηση, το έγγραφο του Μοτρέπου θα γνωρίζετε για τις θετικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις ιδιωτικής Εδώ θέλουμε να υπάρχει σεβασμό των, του Διεθνού δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλε τι περιοχέ ένοπλων σειράξεων. Αυτό το στηρίζουν και ο ΩΣΑ και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σημαντική είναι η κατάργηση τη θανατική ποινή με στρατηγική κοινή με όλους τους προσπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες όπου ενεργοποιούνται, με την αντιμετώπιση των αντιπίνων και με σαφή στήριξη της ε, Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επίσης ε, για τον, ε, για τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών, η Ελβετία γνώρισε κάποιους εμφύλους πολέμους στα 700 χρόνια της ιστορίας της, λιγότερο αιματηρούς από τη, αιματοβαμένους από ό,τι αυτούς της ε, υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η, η δική μας ειρηνική εθνική συνύπαρξη είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και γι' αυτό ακριβώς έχουμε αναπτύξει σε διεθνές, στο διεθνές προσκήνιο τέτοια δράση ώστε τα τελευταία χρόνια να έχουμε φέρει πέρα τουλάχιστον 30 διατησίες ε, Τουρκίας, Αρμενίας, Κολομβίας, Νεπάλ, Σουδάν, Ρωσίας και ούτω καθεξής. Η Ελβετία πιστεύει ότι δεν μπορεί κανείς να αφήσει πίσω το παρελθόν σε μια περίοδο μετά από μια ε, ένοπλη σύραξη, εάν δεν υπάρξει αποκατάσταση και δέσμευση για μια επανάληψη των εχθροπραξιών, καθώς και προστασία των θυμάτων. Ε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κολομβία, όπου δείξαμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε αντιμετωπίζοντας σωστά τα, τις πληγές που έχει αφήσει το παρελθόν. Έχουμε μια σειρά από εμπειρογνώμονες που δραστηριοποιούνται σε κοινέ επιχειρήσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως στο Μαλί και αλλού. Δύο-τρία παραδείγματα επίσης υλοποίησης η Αραβική Άνοιξη. Η Ελβετία αμέσως στην Αίγυπτο προέβλεψε αποστολές ε, στήριξης για την μετάβαση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υπάρξουν οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονταν για την νέα κυβέρνηση και λόγω της Αραβικής Άνοιξης, στήριξη του συστήματος ασφαλείας ώστε το σύστημα ασφάλειας να εξυπηρετεί τα συμπεριόντα του ε, πληθυσμού συνολικά και όχι μόνο μιας κοινωνικής τάξης, μιας πατρίας ή ενός πολιτικού κόμματος. Επίσης στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε γενικές γραμμές όπως με το παράδειγμα τη ε, τηνησιακή τηλεόρασης, του τηλε, μάλλον ραδιοφώνου, του επίσημου φορέα που δεν ήταν πια στα χέρια της εξουσίας, αλλά εξυπηρετούσε όλον τον πληθυσμό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορεί κανείς να εξυπηρετήσει όλα αυτά με μέτρα όπως το πάγωμα των υπηρεσιακών στοιχείων, κάτι που ήδη έχει ε, γίνει, έχει αρχίσει να υλοποιείται μέτρο για περιουσιακά στοιχεία στην Τινησία, στη Λιβύη, στην Τουρκία και στην Αίγυπτο. Ε, ο στόχο είναι να ξεκινήσουν οι κατάλληλε διαδικασίε με τι απαραίτητε προσφυγές και ότι ο καθένα έχει ανακτήσει τα χρηματικά ποσά που το αναλογούσαν προ όφελος ολόκληρου του πληθυσμού. Η Ελβετία λοιπόν παρακολουθεί τι γίνεται στι συγκεκριμένε χώρες με διαδικασίες ώστε την κατάλληλη στιγμή να παρέμβει. Και βεβαιωνόμενοι ότι ε, οι κανόνες έχουν γίνει σεβαστοί και αποδίδονται σωστά τα περιουσιακά στοιχεία εκεί που έπρεπε. Δεύτερο παράδειγμα, η Συρία. Η πολιτική τη Ελβετίας στη Συρία εντοπίζεται σε τρει άξονε. Πρώτον, ο σεβασμός του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έπειτα αυξημένη ανθρωπιστική βοήθεια, 70 ε, δις ευρώ ως τώρα και η αντιμετώπιση των χημικών όπλων. Εδώ μιλάμε για ανθρωπιστική βοήθεια παρέχεται και στις γειτονικές χώρες, στην πράξη δηλαδή επιτόπου, αλλά και με στήριξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή των αντιπολιτευόμενων ομάδων ε, ή του, της κοινωνίας των πολιτών στην ε, Συρία. Ε, η θέση της γυναίκας στην Συρία του σήμερα, η δράση της κοινωνίας των πολιτών είναι κάτι που προσπαθούμε να στηρίξουμε. Ο Αραβικός Σύνδεσμος επίσης με την συνάντηση που προβλέπεται αύριο είναι κάτι στο οποίο παρενεύει η Ελβετία προσπαθώντας να βοηθήσει στη διοργάνωση και προτείνοντας θέματα όπως το πώς μπορεί κανείς να καταλάβει την άλλη πλευρά όταν περνάει σε διάλογο, πώς μπορεί να οργανώσει το διάλογο, η Ελβετία δεν είχε σκοπό να συμμετάσχει αυτή αυτή στι συνομιλίε, απλώ να οργανωθούν οι διαπραγματεύσει για να καταλήξουν στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Επίση, η, καλύτερη, αντιμετώπιση τη ατιμορρησία. εδώ υπήρξε προσφυγή στο Διεθνέ Δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Συρία. Ε, το Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που μας αφήνει ελπίδες ότι με την σύνοδο του Συμβουλίου του αρμόδιου Συμβουλίου του Δικαστηρίου θα υπάρξει και απόδοση ευθυνών. Επίσης για τον ΟΑΣΕ, ε, ένας οργανισμός που υπήρξε θύμα της επιτυχίας του, είναι κάτι που σήμερα επιστρέφει και πάλι στο προσκήνιο για, τον, για την αποφυγή της, ε, των διχασμών στην Ευρώπη Ξέρουμε και είδαμε τι έγινε με την Αρμενία και την Ουκρανία πρόσφατα. Ελπίζουμε λοιπόν τις στενές πολιτικές επαφέ που έχουμε με τη Ρωσία να, την, ε, να τις εκμεταλλευτούμε για να διευκολύνουμε την προσέγγιση σήμερα, δίνοντας έμφαση στα δικαιώματα του ανθρώπου, το σεβασμό της ελευθεροτυπίας, καθώς και την θέση, την τοποθέτηση της Ελβετίας που το νόμο ψηφίστηκε στην Ουκρανία στις 16 Ιανουαρίου. Εδώ Βλέπουμε να υπάρχει βασική διαφορά μεταξύ των χωρών όπου η προοπτική ένταξη είναι ο καλύτερο παράγοντα σταθεροποίηση. Η Ελβετία εδώ θέλει να στηρίξει τι χώρε αυτέ αυτή τη διαδικασία, όπω τα Βαλκάνια. Από την άλλη όμω, στο νότιο Κάφκασο κατά την υπερδινιστερία βλέπουμε ότι οι συνθήκε είναι πολύ πιο δυσχερεί. Εκεί λοιπόν πρέπει να χτίσουμε ξανά γέφυρε επικοινωνία, να χρησιμοποιήσουμε το περιθώρια ε, διαλόγου που, υπάρχει, που υπάρχουν με την Τουρκία, την Αρμενία, τη Γεωργία και τη Ρωσία και να μην υπάρχει πλέον διχασμός στην Ευρώπη. Τώρα για τις διμερείς σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακούσατε τον κύριο David και από τη χθεσινή, David Sullivan και από τη χθεσινή του παρέμβαση ότι είμαστε ο τέταρτος εταίρος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, επενδυτής 1,5 εκατομμύρια καθημερινά συναλλαγές μεταξύ Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερα από ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Μεξικό ή με τον Καναδά. Η Ελβετία λοιπόν είναι ε, ιδιαίτερα δραστήρια ε, στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα εκατομμύριο Ελβετού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του Μπαλίν και ε, εδώ μας ενδιαφέρει να έχουμε ε, απαραίτητη, συνεργασία. Η Ελβετία έχει ψηφίσει πριν από 20 χρόνια όχι στον, ε, στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως υπάρχει μια τομεακή προσέγγιση πλέον, η οποία επέτρεψε να διευρυνθεί η υλοποίηση και ισχύ του ευρωπαϊκού δικαίου και στον ευρωπαϊκό χώρο ε, προς όφελος και των δύο πλευρών. Ε, εδώ να σας δώσω ε, και να σας εξηγήσω ότι εμείς δεν είμαστε απλώς επιλεκτικοί και δύσκολοι. Ε, ο στόχος ήταν να λύσουμε το πρόβλημα που παρουσιάζει η γεωγραφική θέση της χώρας στο μέσον της Υπήρου, στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Υπήρου, αλλά να λύσουμε και άλλα προβλήματα όπως την κυκλοφορία των προσώπων, τα, τις χρυσές ε, και οδικές μεταφορές, ε, την αεροπλοεία, την, τι εμπορικέ συναλλαγέ δεν μπορούσε να μην υπάρχει συνεργασία. Οι εμπορικέ συμφωνίε που έχουν συναυθεί ω τώρα είναι προ όφελο των δύο πλευρών και η μόνη προσέγγιση που θα μπορούσε να Δεχτεί η Ελβετία στις σχέσεις προσέγγισης με την ε, Ένωση δύο άξονες και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να τα δούμε τα πράγματα εκ παραλλήλου με την σταδιακή ανάδυση μιας κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. Όλοι οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί η Ελβετία είναι για να βεβαιωθεί ότι η συνύπαρξη αυτή ε, θα επιτρέψει την εθνική μας ενότητα. Οι Ελβετοί πάντοτε ανησυχούν ότι κάθε δέσμευση για την εξωτερική πολιτική, κάθε δράση στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής μπορεί να φέρει τον διχασμό της χώρας. Η τελευταία στρατιωτική δράση της ε, Ελβετίας ήταν το 1615 στη μάχη του Μαρινιάν και ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα τότε. Ε, οπότε η ανησυχία αυτή δεν είναι πάντοτε εκπεφρασμένη, όμως οι Ελβετοί έχουν πάντοτε αυτό το μέλημα ε, τη θεσμική τους αφοσίωση στο εσωτερικό της χώρας και όχι τόσο σε εξωτερικούς στόχους. Γι' αυτό άλλωστε γίναμε και ήμασταν και μέλη του αργήσαμε να γίνουμε μέλη του ΟΗΕ και η διαδικασία της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς θα είναι ακόμη πιο αργή. Αλλά για τις διασυνοριακές μας ε, ε, ε σχέσεις η Ελβετία βασίζεται σε έναν πολιτικό μηχανισμό, όχι σε ένα έθνο, σε μια γλώσσα. Ο πληθυσμός λοιπόν ε, φαίνεται να απειλείται εάν η Ελβετία συμμετάσχει σε έναν ανώτερο διεθνή οργανισμό αυτό αισθάνονται οι Ελβετοί. Οπότε η Ελβετία θα χρειαστεί καιρό για να βρει τη φωνή τη στο διεθνή φόρα. Όμω αυτό είναι ένα άλλο παράδοξο. Η Ελβρά όπου ο λαό τη ε, αποφαίνεται όλο και πιο συχνά για τις ε, ευρωπαϊκές αποφάσεις, του ευρωπαϊκούς νόμους και το κοινοτικό κεκτημένο. Για την κυκλοφορία των προσώπων, τη διεύρυνση της Ρουμανία, με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, για το Σέγγεν και το Δουβλίνο. Κάθε φορά ο ελβετικός λαός ενέκρινε τις αποφάσεις ε, de facto ενέκριναν τι αποφάσει που έχουν ληφθεί σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και που στη συνέχεια υλοποιήθηκαν και σε εμά. Ε, αντικείμενο διαπραγματεύσεις, όχι διαπραγματεύσει, αλλά προετοιμάζουμε τι διαπραγματεύσει ώστε το Ομοσπονδιακό κράτο να προβλέψει ένα νόμο για να υπάρχει ένα θεσμικό πλώσιο για τι θεμαϊκέ μα σχέσει με την Ένωση. Περιμένουμε την εντολή της Ένωσης, έχετε και εσείς τις εσωτερικές σας συνομιλίες, αλλά οι συνομιλίες σε ελβετικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η Ένωση και σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει να καλύψει τις διαφορές όπως έχει γίνει ως τώρα και εντός ε, της Ένωσης με τα δικά της κράτη-μέλη χωρί σε καμία περίπτωση να κυδεύεται ο αρχικό στόχο. Και ελπίζουμε ότι σε όλα αυτά θα μπορέσει η Ελβετία να βρει τη θέση τη. Και με ένα παράθεμα ε, θα ήθελα να κλείσω λέγοντα ότι η Ελβετία εργάζεται σε κοινού στόχου με την Ένωση στο διεθνέ προσκήνιο. Οπότε για τι αμοιβαίε κοινέ μα σχέσει θα ήθελα να αναφέρω έναν ε, Ελβετό συγγραφέα που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, ο οποίο λέει ότι όταν αφήσαμε τον χώρο το κράτος της κοινωνικής πρόνοιας, αρχίσαμε να υπολογίζουμε τα ωφέλη ε, του καινούριου. Δηλαδή, αυτό που μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα και όχι ο υπολογισμός αυτός καθεαυτός. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάλεγαρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να αποφεληθώ από την ευκαιρία αυτή να σας καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ μέρους της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις μας με την Ελβετία. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι η σχέση μας με τις χώρες ΕΖΕΣ είναι μια πολύ στενή σχέση. Η πιο στενή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες και η Ελβετία είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπατε και εσείς, στον τομέα του εμπορίου αλλά και στον ε, τομέα μετακίνησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, Ελβετία και Τούμπαλιν. Είναι τρίτος ε, οικονομικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετία για τα αγαθά και τις υπηρεσίες μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Έχει ενσωματωθεί πάρα πολύ καλά στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά αλλά και σε άλλες πολιτικές με πάνω από 120 διμερείς συμφωνίες. Εννοείται ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ είναι σημαντικές, όχι μόνο οικονομικά, αλλά Ελβετία εννοεί προφανώς ο μιλητής, εξαιτίας του γεγονός ότι βρισκόμαστε κοντά, ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και έχουμε σημαντικές επαφές μεταξύ των πολιτών μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι ζωτική σημασίας οι σχέσεις μας να βασίζονται σε στέρες θεσμικές βάσεις και πλαίσια. Γιατί έτσι μπορούν να έχουν μεγαλύτερα ωφέλη και οι επιχειρήσεις μας και οι πολίτες μας και σήμερα αλλά και στο μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει τις απόψεις του σε σχέση με τα θεσμικά ζητήματα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ελβετίας με δύο κοινοβουλευτικά ψηφίσματα τα οποία εγκρίθηκαν το 2011 και το 2012. Το μήνυμα κλειδί είναι ότι το μελλοντικό θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τους Ελβετούς πολίτες και επιχειρήσεις. Θα πρέπει η ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων που θέλουν να υποφεληθούν από τις ε, σχέσεις ε, μεταξύ μας, η ζωή τους λοιπόν να είναι πιο εύκολη. Γι' αυτό και χρώμαστε πάρα πολύ για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και για το ότι προσπαθούμε να βρούμε μια λύση σε ό,τι θεσμικά ζητήματα προκύπτουν. Και θέλω να υποφεληθώ από αυτήν την ε, ευκαιρία για να συγχαρώ το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο που ενέκρινε την ελβετική εντολή Ξέρω ότι υπήρξε διαβούλευση όπου κατάφερε η κυβέρνηση να έχει τη στήριξη των βουλευτών, των καντονίων αλλά και των κοινωνικών εταίρων. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για τη δικιά σας προσωπικά τη δράση στη διαδικασία αυτή και ξέρω ότι εσείς και ο κύριος Σάλιβαν συνεργάζεστε στενά. Η ελβετική κυβέρνηση λοιπόν ενέκρινε την εντολή για τις διαπραγματεύσεις το Δεκέμβριο. Ελπίζουμε ότι το ίδιο θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σύντομα και ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις έτσι θα αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παραμείνει δεσμευμένο στους στόχους της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας στο θεσμικό τομέα. Επ' αυτού είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι κάθε συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας θα υποβάλλεται σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη υιοθετήσει τη στάση του εν ώψη της επερχόμενης διαπραγματεύσης. Εμείς πιστεύουμε ότι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας θα πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με την αναβάθμιση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή και της ε, Ομοσπονδιακής Ελβετικής Βουλής. Προτείνω λοιπόν μέσα στο νέο πλαίσιο να συμπεριλάβουμε και έναν διακοινοβουλευτικό πυλώνα ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελβετικό Κοινοβούλιο να μπορούν να συμμετέχουν εκεί με ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας. Έτσι μπορούμε να συνεισφέρουμε θετικά στις εξελίξεις. Και πριν ολοκληρώσω, αν έχετε την ευκαιρία ίσως θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε περισσότερο για το δημοψήφισμα που λαμβάνει η χώρα στις 9 Φεβρουαρίου που είναι κατά της μαζικής μετανάστευσης τι επιπτώσεις θα έχει αν περάσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία. Προσβλέπω λοιπόν στις απαντήσεις σας και γενικότερα στη συζήτηση που θα κάνουμε για τα θεσμικά ζητήματα στην Ελβετία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχετε ήδη ένα ερώτημα. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Άννα Γκάμα, τη συντονίστρια των σοσιαλιστών για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, να λάβει το λόγο για δύο λεπτά, Άννα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Γραμματεύ. Έχω εκτιμήσει ιδιαίτερα την παρέμβασή σας. Θα ήθελα να σας ε, θέσω ένα ερώτημα, πέραν του γεγονότος ότι είπατε πολλά για την ιδιαιτερότητα του ελβετικού χαρακτήρα. Θα ήθελα να σταθώ στη θεσμική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας το θέμα του, της ε, δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δεν θέλει να αποδεχτεί η Ελβετία ως ε, τελικό ε, επιδιαιτητή. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε γιατί. Γιατί φυσικά είναι και ένα πολιτικό θέμα, είναι θέμα το οποίο πρέπει να αποφασίσουν οι ελβετικές αρχές. Ένα άλλο σημείο Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια είναι η θέση της κυβέρνησής σας. Γιατί πιστεύω ότι η κυβέρνησή σας δεν θέλει να γίνει το δημοψήφισμα αυτό για να εδραιώσει ποσοστώσεις μεταναστών. Το δημοψήφισμα αυτό που αναφέρθηκε για τις 9 Φεβρουαρίου που έχει να κάνει με ποσοστώσεις με των μεταναστών. Έχουμε πολλούς Πορτογάλους που εργάζονται στην ε, Ελβετία και έχουν τύχει πολύ καλή υποδοχή, Αλλά αυτό φυσικά είναι και αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητος της ε, Τρόικα που οδηγεί τους Πορτογάλους να ξενιτευτούν στην ε, Ελβετία και σε άλλα μέρη ψάχνοντας για εργασία. Τι γίνεται σε εσά και πώς θεωρείτε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις επιπτώσεις αυτού του δημοψηφίσματος αν νικήσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν ποσοστό. Σε ένα τελευταίο σημείο. Άκουσα αυτά που είπατε για την ε, ανάκτηση στοιχείων ενεργητικού από τις χώρες της Αφρικής και εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειές σας. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι για πολλές από τις χώρες μας η Ελβετία, <clears throat> ιδιαίτερα για την Πορτογαλία, λειτουργεί σαν ένας απέραντος φορολογικός παράδεισος. Στην Πορτογαλία έχουν προταθεί δύο φορές ε, φορολογικές αμνηστίες που θα ευνοήσουν αυτούς οι οποίοι έχουν τα χρήματά τους στην Ελβετία και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους. Το 2012 μέσα στα πλαίσια μια διμερούς συμφωνίας με την Ελβετία ήταν δυνατόν να εντοπίσουμε τα άτομα αυτά. Αλλά η Ελβετία ήθελε να παραμείνουν απόλυτα τα ονόματα αυτών των ανθρώπων. Είναι αυτό αλήθεια και αν ναι, αυτό είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε τη λεύκανση χρημάτων. Ο κύριος Πρέντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και για την ε, παρουσίασή σας κύριε Ρωσιέ. Έχω ένα ερώτημα που έχει να κάνει με αυτά τα οποία είπατε για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για τον ΟΣΑ, τον ΟΑΣΕ, συγγνώμη, συγκεκριμένα την υπερνηστερία. Ο πρόεδρος Ρουμανίας είχε δηλώσει πρόσφατα ότι η Φόρμουλα 5 συν 2 δεν είναι αποτελεσματική και ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Ποια είναι η δική σας αντίδραση, δεδομένου ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε συζητήσει ιδιαίτερα για ορισμένε ενέργειες που έχουν λάβει χώρα στην περιοχή αυτή και υπήρξε και μια πρωτοβουλία των Γκαγκαούζων οι οποίοι ζήτησαν να οργανωθεί ένα δημοψήφισμα τον Φεβρουάριο. Ε, έχετε κάποια απάντηση σε όλα αυτά? ή περιμένετε ότι και μέχρι το τέλος της Προεδρίας σας δεν θα υπάρξει καμία βελτίωση στο θέμα αυτό της υπερνηστερίας. Ευχαριστώ. Ο Σερ Ρόμπερτ Άτκινς. Μας τιμά η παρουσία σας κύριε Υφυπουργέ. Ένα θέμα για το οποίο δεν αναφερθήκατε είναι ο αντίκτυπος της ε, παρουσίας της ε, Ελβετίας στα χρηματοπιστωτικά θέματα διαβάσαμε. ότι κανένας Αμερικανός δεν μπορεί πια να ανοίξει λογαριασμό στην Ελβετία γιατί είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος να φορολογηθεί που καμιά ε, ελβετική τράπεζα δεν θα δεχτεί να συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο. Μήπως όμως θα μπορούσατε να πείτε κάτι για τις πολιτικές επιπτώσεις του να ζητούν οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη-μέλη να αρθεί το τραπεζικό απόρριτο των τραπεζικών εργασιών στην Ελβετία που κατά την άποψη πολλών χωρών πρέπει να τροποποιηθεί. Ξέρω ότι αυτό επηρεάζει και άλλες περιοχές όπως είναι το Λίχτενστάν, η Ανδόρα, τα νησιά της Μάχης. Υπάρχει όμως μια τέτοια κίνηση και εσείς βρισκόσαστε στον κολοφόνα της ε, τραπεζικής ε, δραστηριότητας. Ο, τι θα σήμαινε για σας να γνωρίζουν όλοι τι περνάει μέσα από τις ελβετικές τράπεζες. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να σχολιάσετε για τις πολιτικές συνέπειες που θα προκύψουν για τη χώρα σας. Δύο λεπτά μονάχα χρησιμοποίησα. Ευχαριστώ πολύ, Sir Robert. Η κυρία Γετζετζεύσκα. Το είπα σωστά. Πάντα εκτιμάω το θάρρος αυτού που τολμάει να προφέρει το όνομά μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Ήταν πολύ χρήσιμη, ενδιαφέρουσα και ποτέ δεν υπογραμμίζουμε αρκετά το πόσο σημαντικές, πόσο καρποφόρες και χρήσιμες είναι οι σχέσεις μας με την Ελβετική Συνομοσπονδία. Είναι κάτι που η αντιπροσωπεία μας το γνωρίζει πολύ καλά. Συμμετέχω και εγώ στην αντιπροσωπεία για τις σχέσεις μας με την Ελβετία. Κατόπιν τούτων, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνουμε μηνύματα ότι το αίσθημα αυτό δεν το συμμερίζονται όλοι οι Ελβετοί πολίτες. Και αυτό το λέω κυρίως στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης ατόμων, που είναι ένα ζήτημα όλο και πιο επίμαχο στην Ελβετία. Θέλω να αποφεληθώ λοιπόν από την παρουσία σας εδώ και να σας ρωτήσω για τη δικιά σας αίσθηση σε σχέση με το δημοψήφισμα που πρόκειται να λάβει χώρα στην Ελβετία σχετικά με την μετανάστευση. Το Σύνταγμά σας προβλέπει το δημοψήφισμα και με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε το αποτέλεσμα. Σίγουρα είναι θέμα εσωτερικό του ελβετικού λαού. Όμως είμαι πολύ περίεργη να μας πείτε τη δικιά σας την άποψη, τη ελβετική κυβέρνηση, δηλαδή, σε σχέση με το δημοψήφισμα αυτό. Και τα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι το μόνο που έχει να κάνει με την ελεύθερη διακίνηση. Επίσης αναφερθήκατε στο θέμα της επιλογής. Ότι η Ελβετία δηλαδή παίρνει ό,τι τη συμφέρει και αφήνει ό,τι δεν θέλει. υπάρχουν διάφορες ελευθερίες που διασφαλίζονται από τις συμφωνίες της Ελβετίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, υπηρεσιών, ατόμων και όλες οι άλλες ελευθερίες δεν ε, τίθενται υπό συζήτηση έχουμε την αίσθηση ότι εντάξει τα κεφάλαια υπηρεσίες να κυκλοφορούν ελεύθερα, όμως οι άνθρωποι εκεί αμφισβητείται το ζήτημα. Ποια είναι η θέση της ελβετικής κυβέρνησης επ' αυτού λοιπόν. Ευχαριστούμε κύριο Σβάπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπατε για την ε, Ελβετία και το πώς λειτουργεί η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάθε σεβασμό για τα θέματα αυτά και φυσικά έχουμε και κάθε σεβασμό, αν και επιφυλακτικό, σε σχέση με το δημοψήφισμα της 9ης Φεβρουαρίου. Αλλά και 28 χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφέρονται να κρατήσουν τη συνεργασία τους με την Ελβετία παρά το γεγονός ότι είναι πολύπλοκο το πολιτικό σχήμα το οποίο χρειάζεται να οικοδομηθεί και γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι η βάση της συνεργασίας των κρατών μελών και των πολιτών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βασική αρχή θα πρέπει να είναι ότι όλες οι πλευρές, αν θέλουμε να έχουμε αυτή τη μεγάλη ε, ένωση, όλοι θα πρέπει να μπορούν να συμμεριζόνται τα πλεονεκτήματα αυτής της Ένωσης. Γι' αυτό με κάθε σεβασμό, πάντα σεβόμενοι τις συνταγματικές σας δομές και πρόνοιες, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι ελευθερίες διακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών και δεν είναι για μας κάτι που μπορούμε να διανοηθούμε να χαθούν αυτές οι ευκαιρίες των Ευρωπαίων πολιτών να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Θέλω να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Γκόμε από την Σοσιαλδημοκρατική Ομάδα. Λέει ότι έρχονται οι άνθρωποι στην ε, Ελβετία από την Πορτογαλία λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει, έχουν, έχει δημιουργήσει η Τρόικα. Και βλέπουν εκεί πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές ευκαιρίες που έχουν για την οικονομική ζωή και νομίζω ότι αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να μπορέσει να κρατήσει ανοιχτά τα σύνορά της η Ελβετία έναντι των πολιτών και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κάμπελ Μπένεμαν έχει το λόγο. Είμαι μέλος της αντιπροσωπείας κύριε Υπουργέ και είμαι επίση και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Εμπορίου. Υπήρξε μεγάλη συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού σε σχέση με το θέμα του ελέγχου, των ελέγχων μάλλον, από τις μεταναστευτικές αρχές στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι έχετε κάνει μέχρι τώρα για τα θέματα αυτά. Ξέρω ότι υπάρχουν διασφαλίσεις διμερούς χαρακτήρα και ξέρω ότι μπορείτε να περιορίσετε την ε, μακροχρόνια μετανάστευση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε ένα σύστημα με το οποίο μπορεί να γίνεται ο περιορισμός αυτός από τις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρουμανία και Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι περισσότερο για το τι κάνετε τώρα επί τη βάση των κανόνων αυτών και τι θα αλλάξει, επανέρχεται πάντα αυτό το θέμα, εάν περάσει αυτό το δημοψήφισμα. Αν θα έχετε πολύ μεγαλύτερους περιορισμούς ή θα είσαστε στο ίδιο πλαίσιο και θα ήθελα επίσης να ξέρω ποιο ποσοστό της οικονομίας της ε, Ελβετίας εντάσσεται στην ενία αγορά. Άκουσα να λέτε ότι είστε με τον πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω. Αλλά ποιο είναι το ποσοστό της συμμετοχής σας στην ενία αγορά και μέχρι πού θέλετε να φτάσει αυτό το ποσοστό. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Κύριε Γενική Γραμματέα. Κύριε Γκόμες, Το θέμα του ρόλου του δικαστηρίου δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από την εντολή που υιοθέτησε η Ελβετία. Εφόσον εφαρμόζουμε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει. Δεν αμφισβητείται αυτό το θέμα. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα λεπτό σημείο. Εσείς θεωρείτε ότι πρόκειται για πρακτικό ζήτημα, ενώ ο ρόλος ενός ξένου δικαστηρίου για την Ελβετία είναι θεμελιώδες ζήτημα. Και επανέρχομαι εδώ στη δικιά μας πολιτική κουλτούρα που θέλει ότι να είναι ο πολίτης ο οποίος ελέγχει. Είμαστε ρεπουμπλικάνοι στην Ελβετία, δεν έχουμε αριστοκρατία, αλλιώς θα ήμασταν αυστριακοί. Και οι δικαστές ακριβώς της αριστοκρατίας ήταν πρόβλημα για το σύνταγμα της χώρας. Οπότε είναι θεμελιώδης για μας και καταλαβαίνετε για την Ελβετία οι συμβολισμοί είναι σημαντικοί είναι σαν να σας λέγαμε να πάρετε εσείς στην Πορτογαλία τον βασιλιά της Ισπανίας για αρχηγό του κράτους σας. Καταλαβαίνετε πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα αυτό, όπως θα σας έφυγε και εσάς στο παράδειγμα που έδωσα. Τώρα, θέλω να απαντήσω εδώ μεταξύ άλλων και στην κυρία Γερζιζεύσκα. Η θέση της ελβετικής κυβέρνησης είναι σαφής. Εμείς κάνουμε εκστρατεία η κυβέρνηση. Και εγώ 2.000 ομιλίες έβγαλα. Όχι, δεν είναι θέμα επιλογής του διαλέγουμε ό,τι θέλουμε. Όχι, είναι η διαδικασία που ακολουθούμε στη χώρα και η οποία μας κρατάει χώρα. Έχουμε κοινούς πολιτικούς θεσμούς, ενώ έχουμε πολλές ε, διαφορές. Εμείς δεν έχουμε μια φυσική εθνική ενότητα. Όταν λοιπόν παίρνουμε αποφάσεις σε άλλε χώρες καταλήγει το θέμα στο κοινοβούλιο που αποφασίζει. Σε εμά είναι τα δημοψηφίσματα που αποφασίζουν. Εφτά φορές ψήφισαν οι Ελβετοί για το κεκτημένο και πέντε για την ελεύθερη διακίνηση. Εντάξει, δεν υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχουν κάνει δημοψήφισμα και να πήραν ναι για τέτοια δύσκολα ζητήματα. Οπότε η αίσθηση για το θέμα της ελεύθερης διακίνησης, βλέπετε, και εμείς συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες της Ευρώπης και ξέρουμε και εμείς ότι μπορεί το αύριο να είναι πιο δύσκολο από, το σημερινό, από τη σημερινή κατάσταση. Η Ελβετία είναι μια χώρα στην οποία το ζήτημα καταλήγει σε δημοψήφισμα. Αλλά δεν είναι αλλιώ από ότι είναι σε άλλες χώρε, γιατί και άλλες χώρε τι απασχολεί. Με ρωτήσατε αν απαντήσουν ναι οι Ελβετοί στο δημοψήφισμα, τι θα κάνουμε, δηλαδή υπάρξει περιορισμός της διακίνησης, ε, δεν έχουμε προς το παρόν εναλλακτική λύση. Έτσι και αλλιώς Πολύ θα θέλαμε να διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση και να μην περάσουν οι προτάσεις για περιορισμό της μετανάστευσης όπως προβλέπετε στο δημοψήφισμα. Και προσέξτε, εμείς έχουμε ελεύθερη διακίνηση αγαθών και ατόμων, όχι υπηρεσιών. Δεν ισχύει αυτό που είπατε πριν. Για την τρίτη σας ερώτηση, κυρία Γκόμες, όσον αφορά τους ε, οικονομικούς παραδείσους. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα τεράστιο κόστος και έμεσο και άμεσο. Έτσι συμβαίνει με τις ομοσπονδιακές χώρες και στις ΗΠΑ είναι το ίδιο. Το σύστημά μας είναι τέτοιο όπου στην Ελβετία το κράτος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες από το τραπεζικό σας λογαριασμό. Παρόλα αυτά Εμεί συμμορφωνόμαστε πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρξει κατάχρηση και γι' αυτό και η Ελβετία έκανε μεταρρυθμίσει. Η εντολή διαπραγματεύσεων ήταν έτοιμη στην Ελβετία πολύ πριν από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επέκταση τη ε, οδηγία όσον αφορά την φορολογία των καταθέσεων. Η Ελβετία ακολούθησε μια προσέγγιση που ήταν να ε, συγκεντρώνει τον φόρο και μετά να τον παραδίδει πρέπει να πληρώνουν ενδιαφερόμενοι φυσικά τους φόρους τους και έχουμε πάρα πολλές συμφωνίες που καταλήγουν στο να δίνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ε, χρήματα από φόρους στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Τώρα περνάει το θέμα και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι αυτό η ερώτηση και του Σερ Roberts. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Ελβετία ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και συνεργαζόμαστε. Πήρε χρόνο, συμφωνώ, αλλά τώρα έχουμε μπει στο βλάκι. Αυτό που θέλουμε είναι να καταλήξουμε σε διεθνείς προδιαγραφές. Αναφερθήκατε εσείς στα νησιά της Μάχης, εγώ μπορώ να σας αναφέρω τη Σιγκαπούρη. Συνεπώς, αν πράγματι υπάρχει ε, μια διεθνή στάση, βεβαίως και η Ελβετία θα αποτελεί μέρος. Τότε βεβαίως και η Ελβετία θα συμμετέχει. Αλλάζει η στάση της Ελβετίας τα τελευταία χρόνια. Ενώ τα διάφορα φορολογικά καθεστώτα, ο κώδικας δεντολογίας και τα είναι πράγματα που εξελίσσονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε μια ικανοποιητική λύση και για τις δύο πλευρές. Ρωτήσατε για την υπερνηστερία. Όταν συζητήσαμε ε, με τους Σέρβους, γιατί θέλαμε να κάνουμε μια προεδρία για δύο χρόνια, έτσι ώστε να κρατάει πιο πολύ και όχι μόνο ένα χρόνο. Ελπίζουμε να μην ε, ξεχαστεί, πολλές φορές ξεχνιούνται οι προεδρίες ε, της ΟΑΣΕ πολύ γρήγορα. Ορίσαμε λοιπόν δύο ειδικού απεσταλμένους για τα Βαλκάνια και τον Νότιο Κάφκασο. Ο κύριος Μπακοβίτς είναι ο Σέρβος πρέσβης που θα είναι ο ειδικό απεσταλμένος για την υπερδυνιστερία. Η Σερβία λοιπόν κυρίως μαζί μας θα ηγηθεί των διαδικασιών το 5 συν 2 για μας δεν αμφισβητείται από τίποτα. Το βασικό είναι η θέση της Ρωσίας. Ξέρετε ότι δεν έχει αναγνωρίσει την υπερνηστερία σε αντίθεση με ό,τι έγινε στην γεωργική σύγκρουση. Όλα λοιπόν σταμάτησαν με την απόφαση της Ουκρανίας για την αλλαγή των ορίων στην Συμφωνία Σύνδεσης. Κατά τη γνώμη μου το βασικό είναι να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους Ρώσους, να αποφύγουμε κάθε προηγούμενο, κάθε δεδικασμένο και τη συνέχεια την αναλαμβάνει η Σερβία και κατά τη διάρκεια της δικιάς μας προεδρίας αλλά και του χρόνου. Κύριε Σφαμπ, πιστεύω. Η κυβέρνησή μας έχει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και έχει ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα και τα συνδικάτα. Αυτό καταδείχνει και, καταδείχνει και πάλι ότι υπάρχει μια κοινή κίνηση κομμάτων και συνδικάτων κατά της παγκοσμιοποίησης. Αυτό το χίμα Έχει βοηθήσει βέβαια την Ελβετία πάρα πολύ σε οικονομική πλευρά. Υπάρχουν όμως και άλλες πτυχές αυτή της μορφής παγκοσμιοποίησης που είναι τώρα επιτάπητος. Η Ελβετία όπως ξέρετε έχει κάνει πολλές φορές δημοψηφίσματα για το θέμα αυτό, για την ελευθερία διακίνησης, διακίνησης των ατόμων. Η άποψη της κυβέρνησης της Ελβετίας είναι σαφής και εγώ θα συνεχίσω να κρατώ αυτή την ε, κατεύθυνση. Αν υπάρξει μια αρνητική εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα να απορρίψουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Κύριε Κάμπελ, ρώτατε για τον έλεγχο. Για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τώρα και για την Κροατία, ξέρετε ότι εκεί γίνεται διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχουν όρια και περιορισμοί για αυτούς που μπαίνουν στην Ελβετία. Υπάρχουν περιορισμοί για πολίτες τρίτων χωρών. Εκεί είναι που πρέπει να περάσουν από μια πολύ περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία για να αποδείξουν ό,τι χρειάζεται για να προχωρήσουν η στάση των Ελβετών. Και εδώ θα έλεγα κοιτάξτε την αλλαγή της οδηγίας ελεύθερης διακίνησης των υπηρεσιών που τώρα προχωράει στην Ευρώπη. Οι λύσεις που έχουμε εμείς μοιάζουν πάρα πολύ με τις λύσεις που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί, για να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις που δουλεύουν στην Ελβετία τηρούν τις εθνικές προδιαγραφές για ελάχιστο μισθό κλπ. Είναι ένας μηχανισμός που ισχύει στην Ελβετία, που οδήγησε σε κάποιον εκνευρισμό από τις γείτονες χώρες, αλλά δεν αμφισβητούμε την ελεύθερη διακίνηση, απλώς βάζουμε προϋποθέσεις. Αν πάτε να δουλέψετε σε μια άλλη χώρα, πρέπει να τηρήσετε τον νόμο εκεί. Αν φτιάξετε μια επιχείρηση σε μια άλλη χώρα, ως εργοδότης πρέπει να τηρείτε την νομοθεσία της χώρας στην οποία εγκαθίσταται η επιχείρησή σας. Αν ξέχασα κάποιον, συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι τελείωσα. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Γραμματέα, ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας και είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ευχαριστούμε. Well, colleagues. συνάδελφοι, θα ήθελα να καλωσορίσω ιδιαίτερα την εξοχότητά του, τον Μασούντ Μπαρζάνη, πρόεδρο της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν του κράτους του Ιράκ. Ο πρόεδρος Μπαρζάνη αντιμετωπίζει ίσως την πιο δύσκολη εποχή στην ιστορία του Ιράκ και είναι η παρουσία του εδώ ένα παράδειγμα της ελπίδας που υπάρχει για σταθερότητα στην περιοχή. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν έχει ανοίξει το δρόμο για καλύτερες σχέσεις μεταξύ της ε, ε, κυβέρνηση του Ιράκ, της ομοσπονδιακή κυβέρνησης του Ιράκ και μια σημαντική γειτονική χώρα όπω είναι η Τουρκία και επίσης γνωρίζουμε ότι έχετε δώσει μεγάλη βοήθεια σε ένα όλο, ένα αυξανόμενο αριθμό Σύριων προσφύγων. Θα κάνετε εκλογές τον Απρίλιο του 2014 <clears throat> και ελπίζουμε θα μπορέσει να υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύστημα κατανομής των εξουσιών μεταξύ των περιφερειακών οντοτήτων και της κεντρικής κυβέρνησης του Ιράκ. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις σας για το πώς θα μπορεί να επανέλθει η ασφάλεια και η σταθερότητα στο Ιράκ, να προωθηθεί η συμφιλίωση προς το συμφέρον όλου του λαού του Ιράκ. Και θέλω να πληροφορήσω τους συναδέλφους μου ότι τα αραβικά βρίσκονται στο κανάλι 25 και να σας πληροφορήσω επίσης ότι η εξοχότητά του του κυρίου Μπαρζανή θα πρέπει να αποχωρήσει στις 5 ακριβώς. Γιατί έχει μια άλλη υποχρέωση. Σας καλώ λοιπόν να λάβετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή τη συνάντηση, λέει ο κύριος Μπαζένη. Και θα λάβω το λόγο στα αραβικά. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω και να αποτίσω φόρο την στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και υπάρχει μεγάλη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ιράκ καθώς και των περιφερειακών κυβερνήσεων στο Ιράκ σε όλους τους τομείς και ιδίως <clears throat> σε ό,τι αφορά τα εμπορικά και οικονομικά θέματα. Όπως το γνωρίζετε, υπήρξε μία συμφωνία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης του Ιράκ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελπίδα μας είναι ότι η περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο μέσα σε αυτή τη συμφωνία ώστε να συσφιχθούν ακόμα περισσότερο οι δεσμοί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας και ιδιαίτερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου της περιοχής μας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τώρα την τραγική κατάσταση στην οποία ζει ο κουρδικός λαός. Ο κουρδικός λαός υπέστη πολλά δεινά μετά από πολλές εκστρατείες που έλαβαν χώρα εναντίον του στο Ιράκ. Ήμασταν τα θύματα της χημικής επίθεσης που έπληξε τις γυναίκες και τα παιδιά ιδίως την εποχή του Σαντάμ Χουσέιν, επίσης της εκστρατείας Ανφάλ του 1900 που οδήγησε σε 70.000 αγνοούμενους. Μόνο 4.000 πτώματα βρέθηκαν σε κοινούς τάφους στο νότιο τμήμα του Ιράκ. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ακόμα αγνοούνται και δεν έχουν ευρεθεί τα πτώματά τους ακόμα. Προς το παρόν. Ή μάλλον κατά τη διάρκεια αυτής της ε, εκστατείας εναντίον των Κούρδων 5.000 παιδιά και γυναίκες ε, έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στην Χαλάμπτσα λόγω της, ε, χημικής, της χρήσης χημικών όπλων. Στην περιοχή του Κουρδιστάν <clears throat> έχουμε ακολουθήσει την αρχή της ανεκτικότητος και της αποδοχής όλων των άλλων. όταν έλαβε χώρα το 1991 η εξέγερση του κουρδικού λαού, εμείς δεν θελήσαμε την εκδίκηση. Ούτε και μετά από το 2003 διεκδικήσαμε κάποια εκδίκηση. Ανοίξαμε μια νέα σελίδα, μια λευκή σελίδα αντίθετα και για τους εαυτούς μας και για τους άλλους. αφήσαμε κατά μέρο το παρελθόν και έχουμε αποδηθεί σε μια προσπάθεια να προσπαθήσουμε να καταπραίνουμε τον πόνο και τα βάσανα του λαού μας και να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. σε αυτή την πολιτική ανεκτικότητος η περιοχή του Κουρδιστάν έχει καταφέρει να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο σταθερότητας και ασφάλειας. Ένα μεγάλο μέρος διεθνών επιχειρήσεων από διάφορες χώρες έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή μας και έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις στην ε, περιοχή του Ιρακινού, Κουρδιστάν. Ως παράδειγμα, μπορείτε, μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα για να κατανοήσετε την πρόοδο της περιοχής μας. Πριν από το 2003, το κατακεφαλήνα έπειτα ήταν 500 δολάρια, ενώ τώρα βρίσκεται στα 5.000 δολάρια κατά κεφαλή. Έχει δεκαπλασιαστεί δηλαδή καταβάλουμε προσπάθειες για να μπορέσουμε να θεμελιώσουμε δημοκρατικούς θεσμούς στην περιοχή μας και χρειαζόμαστε γι' αυτό τη βοήθειά σας. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά, μας, τη βοήθειά σας για να εδραιώσουμε αυτούς τους <clears throat> θεσμούς με τρόπο σταθερό, υγιή και σύγχρονο. Χρειαζόμαστε την εμπειρία σας στα θέματα αυτά. Ξέρουμε ότι θα δείξετε αλληλεγγύη με τον κουρδικό λαό για να μπορέσει να ασκήσει τα δικαιώματά του. Θέλουμε από εσά να καταβάλλετε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να γνωριστεί η γενοκτονία που έγινε σε βάρος του κουρδικού λαού. Και ζητούμε από εσά επίσης ζητούμε τη συνεργασία σας <clears throat> για να μπορέσει να υπάρξει μια ειδική αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κουρδικό τμήμα του Ιράκ. Γιατί με την ύπαρξη μιας τέτοιας αντιπροσωπείας θα μπορούμε να έχουμε στενότερους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ της περιοχής μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι ακόμα το οποίο θα θέλαμε. Θα θέλαμε να υποστηρίξετε την πολιτική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο Ιράκ προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης δημοκρατίας και για να εδρεωθεί το Σύνταγμά μας και να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία στο Ιράκ. Δυστυχώς, η τρομοκρατία έχει καταστεί ένα φαινόμενο το οποίο σοβεί σε όλο το πλανήτη μας και απειλεί όλο το πλανήτη μας. <clears throat> Έχουμε πληγεί ιδιαίτερα από την τρομοκρατία, εξακολουθούμε όμως να αγωνιζόμαστε κατά των τρομοκρατών. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον της τρομοκρατίας. Όπως έλεγα λοιπόν προηγουμένως, έχουμε θεσπίσει την αρχή της ανεκτικότητος και της ελευθερίας θρησκευτικού συναισθήματος. Και στην κοινωνία μας η γυναίκα έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο και στην κοινωνία μας και στους θεσμούς μας. Χάρη σε αυτή την πολιτική στην σταθερότητα και την ασφάλεια που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε στην περιοχή του Κουρδιστάν. Έχουμε αυτή τη στιγμή υποδεχτεί 250.000 πρόσφυγες, κυρίως Κούρδους από τη Συρία. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και Άραβες πρόσφυγες και Χριστιανοί πρόσφυγες. Έχουμε υποδεχτεί επίσης 200.000 από τους αδελφούς Άραβες μας από το κέντρο και το νότιο τμήμα του Ιράκ που έχουν έρθει στην περιοχή μας για να βρουν καταφύγιο προσπαθώντας να ξεφύγουν από την τρομοκρατία και την ανασφάλεια στις υπόλοιπες περιοχές του Ιράκ. Στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν υπάρχουν και 10.000 χριστιανικά νοικοκυριά περίπου. Οι οικογένειες αυτές είδαν να προστίθενται σε αυτές και άλλες 25.000 οικογένειες από άλλες περιοχές του Ιράκ που έχουν προσπαθήσει να διαφύγουν τη δρομοκρατία που ασκείται σε άλλες περιοχές του Ιράκ. Επιπλέον έχουμε 15.000 πρόσφυγες από την περιοχή Ανμπάρ η οποία αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Η περιοχή μας λοιπόν έχει γίνει, έχει γίνει καταφύγιο για πολλούς Ιρακινούς από το υπόλοιπο Ιράκ. Παρ' όλα αυτά τα γεγονότα, οι εντάσεις συνεχίζονται, αλλά δεν έχει δοθεί η απαραίτητη διεθνής προσοχή στους πρόσφυγες αυτούς που έχουν καταφύγει στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Δεν είχαμε την ε, ε, απαραίτητη διεθνή βοήθεια που δόθηκε σε πρόσφυγες σε άλλα τμήματα του κόσμου. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε προκλήσεις. Εξακολουθούμε να εφαρμόσουμε πάντα μια πολιτική ειρηνική, μια πολιτική ανοχής και ανεκτικότητας και προσπαθούμε πάντα με τις άλλες ε, περιφέρειες του Ιράκ να έχουμε καλές σχέσεις και να σεβόμαστε το Σύνταγμα του Ιράκ. Όπως σας είπα όμως, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας και την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. <clears throat> Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ. Είμαι βέβαιος ότι οι κλήσεις σας θα εισακουστούν. Να καλέσω τώρα τους συναδέλφους να θέσουν τις ερωτήσεις τους ή να σχολιάσουν. Όμως, μια παράκληση. Προσπαθήστε να περιοριστείτε σε 1,5 λεπτό ο καθένας. Διότι, όπως είπα, θα πρέπει να φύγει η εξοχότητά του στις 5 ακριβώς. Η κυρία Γκόμες πρώτη, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Μεγάλη μας χαρά να σας βλέπουμε εδώ, πρόεδρε Μπαζάνη. Και εσείς με υποδεχτήκατε το 2008 όταν ετοίμαζα την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για το Ιράκ. Και έβλεπα ήδη τότε ότι υπάρχει ένα άλλο Ιράκ στη δική σας την περιοχή. Ένα Ιράκ ασφαλέστερο και πιο ανεπτυγμένο. Εδώ εκτιμώ το ρόλο που παίξατε εσείς την ε, περιφερειακή σας, με την περιφερειακή σας κυβέρνηση και συντελέσατε στην ενότητα του Ιράκ. Πιστεύω, επισκεπτόμενοι την περιοχή σας, ότι και εμείς μπορούμε να καταλάβουμε τι διωγμούς και τι γενοκτονίες έχετε υποστεί. Αυτό το ανέφερα και στην έκθεσή μου από τότε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα και μπορούν να γίνουν περισσότερα. Πέραν αυτών έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, λαμβάνω ειδήσει οι οποίες με ανησυχούν. Εδώ και μήνες, εδώ και κάποιους μήνες, λέγεται για το σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λέτε κι εσείς ότι χρειάζεστε την ε, στήριξή μας για την σωστή διακυβέρνηση, αλλά οι ειδήσει που λαμβάνω εγώ λένε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ε, περιοχή με τον δημοσιογράφο που εξέθεσε φαινόμενα διαφθορά διαφθοράς και άλλου είδους προβλήματα, εγκλήματα κατά γυναικών. Κάτι που από τότε το είχαμε εντοπίσει, αλλά για το οποίο δεν έχουν γίνει και πολλά. Η η ε, άλλη με ερώτηση έχει να κάνει με το κίνημα Γκίλαν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τους Κούρδους σε όλη την Τουρκία. Και ποια είναι η άποψή σας για το ενωμένο Ιράκ, για το ενιαίο Ιράκ, εφόσον θεωρήσουμε ότι μπορεί να υπάρχει εξάπλωση του πολέμου και επιπτώσεις και για τις γειτονικές χώρες και για τη δική σας προσωπική κυβέρνηση και όλο το Ιράκ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριο Στίβενσον, πρόεδρο τη Αντιπροσωπεία για τι σχέσει με το Ιράκ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε και πρόεδρε Μπατζανή, είστε πάντοτε ευπρόσδεκτο εδώ. Έχω επισκεφθεί επανειλημμένο στο Κουρδιστάν και την τελευταία φορά είχα την τιμή να σα συναντήσω τον Νοέμβριο τη περσινή χρονιά στο Κουρδιστάν. Επισκέφτηκα τότε κάποιους από τους καταπλησμούς προσφύγων όπου έχουν ε, τοποθετηθεί οι Σύριοι πρόσφυγες. Πρέπει να ευχαριστήσω εσάς και την προσωρινή σας κυβέρνηση για τη δουλειά που κάνετε για την ε, προστασία των προσφύγων. Το είπατε και στην παρουσίασή σας, όχι μόνο με τις εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων από το υπόλοιπο Ιράκ, από τις καταπιεσμένες μειονότητες, ιδίως τους χριστιανούς της χώρας, τους, στους οποίους έχετε παράσχει προστασία, αλλά πραγματικά πλέον διεθνώς αναγνωρίζεστε ως ένας ασφαλής λιμένας και οι Σύριοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό. Θα πρέπει να σας προσφέρουμε περισσότερη βοήθεια και σημειώνω το πολύ σαφές σας μήνυμα. Επίσης θα συμφωνήσω με την κυρία Γκόμες. Πρέπει να στηρίξουμε και εσάς και την έκκλησή σας για την ε, αναγνώριση της γενοκτονίας του Άνφαλ. Επίσης, όπως μόλις είπατε, θα πρέπει να υπάρξει και παρουσία καθώς και δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τόση δυνατότητα ανάπτυξης και άνθησης στην περίπτωση του Κουρδιστάν. Δεν αρκεί μόνο η αντιπροσωπεία μας στη Βαγδάτη. Έχετε, θα έχετε από μας όλη τη στήριξη που χρειάζεστε και την αναγνώριση, κυρία Μπαρζάνη. Ευχαριστούμε, ο κύριος Πέτερινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη μου εκτίμηση κύριε Μπατσάνη για αυτά που κάνετε για το Βόρειο Ιράκ και το Κουρδιστάν, το κουρδικό Ιράν. Ήμουν πριν από τρία χρόνια στο Έρμπιλ όπου υπήρχε μια μεγάλη καθολική εκκλησία και εντυπωσιάστηκα με την ευκαιρία αυτή που είχα να δω ότι μπορούν οι χριστιανοί να ασκούν την θρησκευτική τους λατρεία στο Έρμπιλ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για άλλες χώρες της περιοχής. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το παράδειγμα. Σας είχα συναντήσει και στην Ευρώπη, στο Βερολίνο και είχα εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από εσάς. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα. Πρώτον, ποιες δυνατότητε βλέπετε εσείς για την ε, περιοχή σας για να μπορέσετε να συμβάλλετε στην ε, ευημερία και την ασφάλεια του Ιράκ και της Συρίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω με μεγάλη εκτίμηση τα δύο αυτά ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φαντάλεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας από πλευράς των φιλελεύθερων. Μπορώ να πω ότι σεβόμαστε το γεγονός πως εσείς κάνατε ασφαλή λιμένα για πρόσφυγες στο Ιρακινό Κουρδιστάν και για τον δικό σας το λόγο. Έχω όμως κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, η οριοθέτηση των συνόρων μέσα στο Ιράκ, ανάμεσα στη κουρδική περιφέρεια και την υπόλοιπη χώρα, από όσο ξέρω δεν έχει γίνει. Ποια είναι η κατάσταση, θα γίνει με ειρηνικό τρόπο από πλευράς της κεντρικής Ιρακινής κυβέρνησης. Δεύτερον, πώς βλέπετε να υπάρχει διακανονισμός για τη Σερία. Εμείς δηλαδή ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι νομίζετε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φανόρδεν τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και καλωσορίζω και εγώ εδώ τον ε, κύριο Μπαρζάνη. Πρώτη ερώτηση. Πώς χαρακτηρίζετε την κατάσταση ασφάλειας στην κορδική περιφέρεια του Ιράκ. Αλκαΐντα, ε, ΠΚΚ, υπάρχουν. Δεύτερο, μπορείτε να πείτε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ακόμα όσον αφορά την παραγωγή πετρελαίου και εξαγωγή πετρελαίου. Και τρίτον, που είναι ένα ευρύτερο βέβαια ζήτημα, πώς βλέπετε να γίνονται αλλαγέ στην ε, γεωπολιτική κατάσταση της περιοχής τα επόμενα χρόνια. Προβλέπετε η κορδική περιφέρεια του Ιράκ να γίνει πιο αυτόνομη. Προβλέπετε πιο στενές σχέσεις με την Τουρκία. Αναμένετε αλλαγές στην Βαγδάτη που θα σας έδινε μεγαλύτερα ευχαίρεια κίνησης, δικαιώματα κτλ. Κύριος Πασμακέρ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, εδώ είμαι. Και εγώ με τη σειρά μου σας καλωσορίζω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να ξέρετε ότι είμαστε από αυτού που παρακολουθούμε πολύ καλά την κατάσταση και υποστηρίζουμε τα δικαιώματα για όλους τους λαούς και για τον κουρδικό λαό. Αναφερθήκατε στην τραγική ιστορία. Πράγματι, τώρα έχετε αυτόνομες δημοκρατικές αρχές για τις οποίες σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Λέτε ότι υποδέχεστε και πρόσφυγες και σωστά λέτε ότι θα έπρεπε να σας στηρίξουμε περισσότερο. Ζητήσατε επίσης και αναγνώριση της γενοκτονίας. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την περιφερειακή κατάσταση, στην ε, Συρία από το 2007 η περιφερειακή κυβέρνηση στρέφεται περισσότερο στην Τουρκία. Δίνει περισσότερα οικονομικά κίνητρα. Η κεντρική κυβέρνηση όμως ε, Βαγδάτ και Τουρκίας καταπολεμούν μαζί τον ε, Ασάντ στη Συρία και το Ιράν. Η σχέση σας με την κυβέρνηση της Άγκυρας δοκιμάζεται. Έπειτα, η κατάσταση στη Συρία τι επιπτώσεις έχει στη δικιά σας θέση στην περιοχή. Αποδυναμώνεται αν, ε, σε σχέση μάλλον με το κύρος της κεντρικής κυβέρνησης στη Βαγδάτη. Ο κύριος Σόλτς τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Μπαζανή για τις δηλώσεις σας. Εδώ είμαι. και εμείς παρακολουθούμε από πολύ κοντά την εξέλιξη της κουρδικής αυτονομίας στη δημοκρατία του Ιράκ και η δηλώσει σας ότι υπήρξε μια θετική εξέλιξη στην περιοχή αυτή, σε μια περιοχή πολύπλοκων ε, εθνοτικών ομάδων, εντυπωσιακή. Εσείς μιλάτε για την παρουσία ξένων επιχειρήσεων στην περιοχή σας. Πώς έχει συμβάλει αυτό στο να υπάρξει μια θετική κοινωνική και οικονομική εξέλιξη του Ιράκ και μπόρεσε τελικά να συμβάλει για το σύνολο του Ιράκ. Πόσο υπάρχει λοιπόν υπάρχει συμμετοχή αυτών των ε, εξελίξεων για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που υπάρχουν σε επίπεδο ασφάλειας στην ε, χώρα σας. Παρουσιάσατε το θέμα των περιφερειακών, των τοπικών συνθήκων ασφάλειας για τους Κούρδους. Όταν πρόκειται για τους Κούρδους οι οποίοι βρίσκονται στο Ιράκ, στο Ιράν, στην Τουρκία, στη Συρία, πώς μπορεί το σύνολο του κουρδικού πληθυσμού εκεί να βοηθήσει τη σταθεροποίηση της κατάστασης σε άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη το θέμα το οικονομικό. Η δημιουργία πετρελαιαγωγού από την περιοχή σας προς την Τουρκία. Πόσο έχει συμβάλει σε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Τρεις ακόμα ομίλητες. Πέτρελε, Τάνοκ και Κέλλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος, διότι λίγο πολύ θα επαναλάβω προηγούμενη ερώτηση. Ε, με ενδιαφέρει πολύ η δική σας η θεώρηση μιας συνολικότερης λύσης του κουρδικού εντός της γεωγραφικής ζώνης. Τι άποψη έχετε. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ε, θερμό καλωσόρισμα και από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Εγώ πάντοτε ε, θαύμαζα την δημοκρατία που χτίζεται στο Βόρειο Ιράκ τόσο διαφορετική από τον ταραχώδη Νότο με ευημερία και σταθερότητα και ειρήνη. Βεβαίω με την εκστρατεία Άνφα υπήρξε πραγματική αιματοχυσία και χάθηκαν πολλές ανθρώπινες ζωές και επίσης πρέπει να πω ότι για τους ε, χριστιανούς από τη Συρία προσφέρατε πραγματικά θαυμαστή βοήθεια και σας ευχαριστούμε ξανά γι' αυτό. Τώρα, για το προηγούμενο δημοψήφισμα, ξέρουμε ότι είναι πολύ ευαίσθητο το ζήτημα αυτό, αλλά είναι κάτι που πρέπει να λυθεί. Και ήθελα να μας πείτε τι σχέσεις βλέπετε να διαμορφώνονται με την Τουρκία, ιδίω λόγω του προβλεπόμενου και προγραμματιζόμενου αγωγού. Εδώ να σας συγχαρώ μάλιστα για το νέο αυτό αγωγό, αλλά φαίνεται ότι ενδεχομένως να βελτιώσει και τις σχέσεις με την Άγκυρα. Μπορείτε να το σχολιάσετε. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ, ο κύριος Κελάμ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Απλώς να ενώσω και εγώ τα καλωσορίσματά μου με αυτά των συναδέλφων. Ένα θερμό καλωσόρισμα γιατί πραγματικά το αξίζεται. Η νέα κυβέρνηση έδειξε ότι μπορεί να γίνει κάτι καλό ε, και να υπάρξει αλλαγή με επικοδομητικό και θετικό τρόπο. Το ερώτημά μου είναι ποια η άποψή σας για τις επερχόμενες εκλογές, τις βουλευτικές εκλογές στο Ιράκ. Θα συμμετάσχετε. Τι άποψη έχετε και τι προοπτικές ε, κυβερνητικές βλέπετε να υπάρχουν. Και επίσης μπορείτε να διευκρινίσετε τι είδους βοήθεια χρειάζεστε πρωτίστως. Τρίτον, για τον ε, πετρελαγωγό μιλήσαμε ήδη περιμένετε να υπάρξει κάποια συμφωνία με την κυβέρνηση της Βαγδάτης, ε, κάποια συμφωνία για την ε, κατανομή των πόρων. Πώς βλέπετε στο μέλλον διαμορφώνονται οι εξαγωγές πετρελαίου και πώς θα μοιράσετε ουσιαστικά το πετρέλαιο, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα πραγματικά ακροτελεύτιος ε, παρεμβαίνων ο κύριος Μπέλτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Σας χαιρετίζω. Πολλές φορές είχα την ευκαιρία να βρεθώ στο Βόρειο Ιράκ. Μια ερώτηση. Ως προτεστάντης χριστιανός, με ενδιαφέρει η κατάσταση της χριστιανικής κοινότητας, της μειονότητας της χριστιανικής που βρίσκεται εκεί. Εσείς πιστεύετε ότι εντάσσετε καλά. Εγώ έχω ακούσει ότι πάνε δυτικά και ότι τελικά το Ιράκ θα καταλήξει να είναι χωρίς χριστιανούς. Κάτι πολύ θλιβερό για την ε, χριστιανική κουλτούρα. ποια είναι η κατάσταση με την χριστιανική μειονότητα και την χριστιανική εκκλησία στο Κουρδιστάν. Μ' ακούω δυσάρεστα νέα από εκεί, ελπίζω εσείς να με καθισχάσετε. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Τώρα, πολλές οι ερωτήσεις. Αυτό δείχνει πόσο πολύ μας ενδιαφέρει το θέμα και πόσο πολύ εκτιμάμε το δικό σας το έργο εκεί. Παρακαλώ, για να απαντήσετε. Και μην ξεχνάτε ότι έχετε και αεροπλάνο, ε? την πτήση σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα θέματα και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Στην πρώτη ερώτηση καταρχήν της κυρίας Γκόμες. Θέλουμε να οικοδομήσουμε θεσμούς. Το έχουμε ξεκινήσει διατηρώντας την ελευθερία μας γιατί κάθε πολίτης της περιφέρειας του Κουρδιστάν είναι ελεύθερος για τις επιλογές του όσον αφορά την ε, θρησκεία του, τις πολιτιστικές του συνήθειες κλπ. Φυσικά και υπήρξαν απειλές. Είναι μία παραβίαση όμως αυτή που εμείς καταδικάζουμε. Συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, δυστυχώς, τακτικά. Εμείς όμως προσπαθούμε να τα καταπολεμήσουμε. Πρόκειται για παραβιάσεις. Όσοι είναι πεπισμένοι για... Μάλλον, εκείνοι για τους οποίους ξέρουμε ότι πράγματι προχώρησαν σε τέτοιου είδους παραβιάσεις και κλίματα, τιμωρούνται όπως πρέπει. Επίσης, για άλλε ερωτήσεις που κάνανε πολλοί από εσά, οπότε θα προσπαθήσω κάπως συγκεντρωτικά να απαντήσω. Σύρια. Η κατάσταση εκεί είναι βέβαια ιδιαίτερα ανησυχητική για μας. Για ολόκληρο το Ιράκ πρώτα απ' όλα, αλλά και για την κουρδική περιφέρεια. Όλος ιδιαίτερος. Όλα όσα συμβαίνουν στη Συρία έχουν άμεσα επιπτώσεις στη δικιά μας χώρα. Μετά από έξι χρόνια σταθερότητας, στις 26 Σεπτεμβρίου που μας πέρασε στο Ερμπίλ είχαμε τρομοκρατική επίθεση. Και οι υπεύθυνοι που έρχονται από τη Συρία μας ανησυχεί λοιπόν η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια της χώρας μας. Τι εναλλακτική υπάρχει. Υπάρχουν ε, διαφορετικές οργανώσεις, ε, γκρουπούσκουλα, τρομοκρατικές οργανώσεις που εμφανίστηκαν και που δραστηριοποιούνται στην Συρία. Υπάρχει η ΓΑΕΣ που είναι το Ισλαμικό κράτος, υπάρχει το ELL και διάφορες άλλες μικρές ομάδες που πρόσκειται στην Αλκαϊδά. Τρομοκρατικές οργανώσεις που αποτελούν βέβαια απειλή για ολόκληρο το Κουρδιστάν. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει με τίποτα να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτές τις ε, ομάδες να έρθουν πιο κοντά στην εξουσία στο Ιράκ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις φαγές που γίνονται σε βάρος αθών πολιτών και αμάχων. Γι' αυτό η διάσκεψη της Γενέβης θα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι έτσι ο λαός της Συρίας θα μπορέσει να αποφασίσει για το μέλλον του. Δεν λέω ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. ούτε ότι έχω πάρα πολλές προσδοκίες από την Γενέβη 2. Εμείς προσφέραμε ό,τι βοήθεια μπορούσαμε, ανθρωπιστική βοήθεια καταρχήν, προς τους Σύριους αδερφούς μας. Αυτοί που φτάσανε δηλαδή στο Κουρδιστάν του Ιράκ τους υποδεχτήκαμε και τους βοηθήσαμε. Το οφείλουμε αυτό γιατί πρόκειται για αδερφούς μας. Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις του Ιράκ με τη Συρία. Ο φόβος, αυτός τον οποίο αναφέρθηκα πριν, το νιώθει κάθε πολίτης. Ποια είναι η εναλλακτική. Προς το παρόν δεν είναι προφανές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι δημοκρατικές δυνάμεις ή ότι ελεύθερος ο στρατός της Συρίας θα είναι η εναλλακτική λύση για να αναλάβει την εξουσία στη χώρα. Γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν μερικές φορές το πάνω χέρι και βρίσκονται στα σύνορά μας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε οργανώσεις που πρόσκειται στην Αλκαΐδα να δραστηριοποιούνται στα σύνορά μας. Αυτή είναι μια απειλή απευθείας για την περιφερειά μας. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Αυτό που μπορούμε πάντως να πούμε είναι ότι ευχόμαστε από βάθους καρδίας οι Σύριοι να μπορέσουν να αποφασίσουν για το μέλλον τους μακρά από κάθε τρομοκρατική επιρροή. Μια άλλη ερώτηση που μου τέθηκε είναι η οριοθέτηση των εσωτερικών συνόρων στο Ιράκ ανάμεσα στην δικιά μας περιφέρεια και το υπόλοιπο Ιράκ. Ποια είναι η άποψη της κεντρικής κυβέρνησης. Το άρθρο 140 του συντάγματος προβλέπει εξομάλυνση της κατάστασης στις περιφέρειες όπου υπήρξαν δημογραφικές αλλαγές, το Κυρκού και αλλού δηλαδή. Στη συνέχεια πρέπει να υπάρξει απογραφή και μετά την απογραφή πρέπει να προβλέψουμε δημοψήφισμα. Όταν εμείς δηλώσαμε πως συμφωνούμε με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δεν είχαμε ψευδεστήσεις για την άποψη του Κυρκούκ, που είναι κουρδική πόλη, όπου κύρια εθνότητα δηλαδή είναι οι Κούρδοι. Το άρθρο λοιπόν 140 αργήσαμε να το εφαρμόσουμε, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση. Δεν είπαμε ότι η πόλη αυτή ή ότι η περιφέρεια αυτή πρέπει να ενταχθεί στο Κουρδιστάν. Αφήνουμε ελεύθερο το λαό, τους κατοίκους να αποφασίσουν. Θέλουμε όντω να εφαρμοστεί το άρθρο 140 του συντάγματο, Άρθρο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής αυτής να ε, διαθέσουν τον εαυτό τους όπω θέλουν. Αυτοδιάθεση δηλαδή. Έχουν τη δυνατότητα για αυτοδιάθεση, αν το αποφασίσουν. Τώρα μου ζητάτε να περιγράψω την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στο Κουρδιστάν να πω τη γνώμη για την παρουσία της Αλκάιντα, του ΠΚΚ, τρελαϊκές εξαγωγές κτλ. Πρώτα απ' όλα, δούμε την κατάσταση ασφάλειας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η ασφάλεια στο Κουρδιστάν υπάρχει 100% πουθενά εξάλλου. Αλλά νομίζω ότι οι τρομοκράτες δεν μπορούν να έχουν βάση στο Κουρδιστάν. Μπορεί βέβαια να μπουν από άλλες περιοχές, Μοσούλ, Κυρκούκ ή άλλη πόλη, αλλά να διατηρούν μόνιμη βάση στο Κουρδιστάν, αυτό είναι στην πράξη αδύνατο. Σίγουρα εισχωρούν στο έδαφος από άλλα σημεία στις 29 Ιουλίου για παράδειγμα έγινε αυτό. Δεν είναι όμως βάση τους, τρομοκρατική βάση. Συγκρίνοντας με άλλες περιφέρειες του Ιράκ ή άλλων χωρών, μπορούμε να πούμε με αρκετή βεβαιότητα ότι η κατάσταση στο Κουρδιστάν όσον αφορά την ασφάλεια είναι ικανοποιητική. Αντιστεκόμαστε και υπάρχουν δεκάδες και εκατοντάδες ε, ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Κουρδιστάν. Απόδειξη δηλαδή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα για την οποία σας μίλησα πριν. Η Ελκαΐντα δεν έχει μόνιμη βάση στο Κουρδιστάν. Μπορεί να εισχωρήσει. Πεκακά τώρα είναι παρόντες στα σύνορα. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου το Κουρδικό Κόμμα Εργαζομένων να μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία με την τουρκική κυβέρνηση. Η πολιτική διαδικασία πάει ένα βήμα μπρος ένα πίσω, αλλά έχει μπει στη, στο αυλάκι και εμείς θα κάνουμε ό,τι προσπάθειες μπορούμε από τη δικιά μας την πλευρά για να συνεισφέρουμε στην επιτυχία της διαδικασίας αυτής. Εξαγωγές πετρελαίου τώρα. Το Σύνταγμα, το Ιρακινό Σύνταγμα, μας επιτρέπει να εξάγουμε το πετρέλαιό μας. Οι σχετικές διατάξεις στο Σύνταγμα προβλέπουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο ανήκουν στον κουρδικό λαό. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και το επόμενο στον Ιρακινό λαό, συγγνώμη. Και το επόμενο εδάφιο λέει ότι οι περιφέρειες στις οποίες το έδαφος βρίσκεται το πετρέλαιο έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τα πετρελαϊκά αποθέματα σε συνεννόηση με την κεντρική κυβέρνηση. Υπάρχει ένας νόμος, τον οποίο υπογράψαμε, εγώ ίδιος και ο Πρωθυπουργό το 2007, που είναι παράρτημα στην νομοθεσία, που λέει το παράρτημα ότι αν δεν περάσει ο νόμος, τότε η κεντρική κυβέρνηση και η περιφέρεια του Κουρδιστάν έχουν δικαίωμα να συνάψουν συμβάσεις με πετρελαϊκές επιχειρήσεις μέχρι να εγκριθεί τελικά ο νόμος. Προς το παρόν λοιπόν τηρούμε τις διατάξεις του συντάγματος και συγχρόνως έχουμε διαπιστώσει ότι φτιάχνεται αγωγός στην τουρκική επικράτεια. Πριν από δύο μέρες μάλιστα μία αντιπροσωπεία με τον Πρωθυπουργό πήγανε στη Βαγδάτη για να συζητήσουν το θέμα αυτό. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέχρι να καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δράσεις μας εγγράφονται πλήρως στα πλαίσια του συντάγματος το οποίο τηρούμε απόλυτα. Δεν πρόκειται να παρετηθούμε από τα σταγματικά μας δικαιώματα. Τώρα η γεωγραφία θα αλλάξει μετά από την σημερινή κατάσταση. Στρεφόμενοι προς το μέλλον, λοιπόν, θα λέγω ότι σε 20 χρόνια θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Πώς θα έχουν αλλάξει, αυτό δεν μπορώ να το πω, γιατί δεν μπορώ να μαντέψω. Όσον αφορά όμως την κατάσταση, στην περιφέρεια του Κουρδιστάν. Πρέπει να σας πω κυρίες και κύριοι ότι το Κουρδιστάν έχει τα ίδια δικαιώματα όπως και τα άλλα έθνη και οι άλλοι οι λαοί με τους οποίους συνεπάρχουμε στην περιοχή. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτά από τα οποία χαίρουν οι άλλοι λαοί στην περιοχή. Εμείς δεν ζητήσαμε τη γνώμη του κουρδικού λαού για να ξέρουμε αν θέλει να είναι ανεξάρτητο, αυτόνομο ή όχι, η πραγματικότητα είναι σκληρή, είναι πικρή και το δικαίωμα του κουρδικού λαού για ανεξαρτησία θα προχωρήσει όχι όμως με τη βία, αλλά ειρηνικά, με διάλογο και συμφιλίωση. Θα πάρει όσο χρόνο χρειαστεί γιατί είναι ένα θέμα το οποίο με τίποτα δεν μπορεί να διευθετηθεί με βία και όπλα. Είναι όμως ένα απόλυτα θεμητό δικαίωμα και θα πρέπει να τηρηθεί. Όπως είπα και πριν, θα τηρηθεί. Το δικαίωμα αυτό δηλαδή θα το κερδίσουμε ειρηνικά. Όσον αφορά τώρα τις επιθέσεις στη Βαγδάτη. Εδώ πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση στις διάφορες περιφέρειες του Ιράκ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η τρομοκρατία είναι μια πραγματικότητα, το βλέπουμε. Τώρα για την καταπολέμηση ακριβώς της τρομοκρατίας πρέπει να σας πω ότι δεν διαφωνούμε καθόλου με την Βαγδάτη. Θα συνεργαστούμε με την Βαγδάτη στον τομέα αυτό περιμένουμε τις επόμενες εκλογές, τις 30 Απριλίου δηλαδή, και ελπίζουμε ότι οι εκλογές αυτές θα οδηγήσουν σε νέα δεδομένα στο Ιράκ και θα μπορέσουμε έτσι να λύσουμε τα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα. Στη δικιά μας την περιφέρεια του Κουρδιστάν θα κάνουμε ό,τι προσπάθειες μπορούμε για να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα αυτά. Η αυτόνομη κυβέρνηση προσεγγίζει στην Τουρκία για οικονομικούς λόγους. Είναι γεγονός, είναι αλήθεια, πως είναι μια όθηση για τις σχέσεις μας με την Τουρκία, που δεν είναι όμως σε βάρος κανένας άλλου. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτές οι σχέσεις που ενισχύονται με την Τουρκία θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή. Είναι καλό λοιπόν να ενισχυθούν οι σχέσεις της περιφέρειας του Κουρδιστάν με την Τουρκία. Αυτό στηρίζει την ειρήνη, είναι υπέρ της ειρήνης. Υπήρξε και μια ερώτηση για τη Σύρια, αλλά νομίζω ότι την απάντησα νωρίτερα. Ρωτάτε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στη λύση των προβλημάτων ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι άλλες περιοχές του Ιράκ. Από την αρχή εμείς στηρίξαμε την Ιρακινή κεντρική κυβέρνηση στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας και επανειλημμένα είπα ότι η δικιά μας η περιφέρεια θα μπορούσε να συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις αυτού του είδους στα σύνορα ανάμεσα στην ε, περιοχή μας και τη Συρία, στη Μοσούλ δηλαδή. Κατά τη γνώμη μου όμως, τα προβλήματα δεν θα λυθούν μόνο με τη βία. Χρειάζεται και πολιτική μεταρρύθμιση και οικονομική μεταρρύθμιση, όπως και κοινωνική. Πρέπει να υπάρξει εθνική συμφιλίωση. Και αυτό πετύχαμε εμείς στη δικιά μας αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν. Εμείς οι Κούρδοι είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τη Βαγδάτη στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας με κάθε δυνατό τρόπο. Πώς θα μπορούσαν οι Κούρδοι να παίξουν κάποιο ρόλο στην περιοχή σε σχέση με τη Συρία, το Ιράν και την Τουρκία. Εμείς θέλουμε τα σύνορα μεταξύ των χωρών αυτών να είναι όπως τα σύνορα που έχετε εδώ στην Ευρώπη, ανάμεσα ας πούμε στη Γαλλία και το Βέλγιο. Μακάρι. Και αυτό όχι μόνο προς όφελος του κουρδικού λαού, αλλά όλων των λόγων της περιοχής. Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ευρώπης και να καταργήσουμε τα σύνορα. Θα ήταν καλό όλες οι χώρες της περιοχής να εμπνευστούν από το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Δεν είναι καλό οι χώρες της περιοχής να συνεχίζουν αυτήν την πολιτική εξωστρακισμού, ομφαλοσκόπησης, ουσιαστικά να εμποδίζουν τους ανθρώπους να κινούνται ελεύθερα από τη μία περιοχή στην άλλη. Αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα σύνορα με ε, στρατιωτικό τρόπο, με στρατιωτική επέμβαση. Το παρελθόν είναι αυτό που είναι, αλλά η κληρονομιά εξελίσσεται. Οι Κούρδοι των διαφόρων χωρών αλλάζουν τις σχέσεις μεταξύ τους, όπως επίσης αλλάζουν και οι σχέσεις ανάμεσα στους Κούρδους και άλλες χώρες. Είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτό. Όσον αφορά τώρα το δικό μου όραμα, πώς βλέπω εγώ τη λύση του Κουρδικού σε ολόκληρη την περιοχή. Πιστεύω ότι η λύση είναι το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Το δικαίωμα δηλαδή να μπορούν οι Κούρδοι να έχουν τη χώρα τους. Όχι όμως με τη βία, όχι με τα όπλα, αλλά με διάλογο. Πιστεύω ότι θα με δικαιώσει το μέλλον και ότι η ευχή αυτή θα γίνει πραγματικότητα κάποια μέρα. Υπήρχαν χώρες που δεν θέλαν καν να ακούσουν τη λέξη Κουρδιστάν. Το γεγονός ότι οι Κούρδοι έχουν δικαιώματα δεν σημαίνει ότι πλήττονται τα δικαιώματα των άλλων. Καθόλου. Αλλά το να μείνει το ζήτημα του Κουρδιστάν χωρίς λύση δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορεί τότε να υπάρχει σταθερότητα ούτε για τους Κούρδους, ούτε για τις χώρες όπου υπάρχει παρουσία Κούρδων. Με ρωτήσατε επίσης κάτι και για την θέση μου όσον αφορά τις επερχόμενες εκλογές. Οι εκλογές αυτές θα λάβουν χώρα στις 30 Απριλίου όπως σας είπα και οι Κούρδοι θα συμμετάσχουν. Χωρίς καμία αφιβολία. Εξάλλου έχουμε και εμείς ε, ψηφοδέλτιο με υποψηφίους που το υποβάλαμε. Από τα αποτελέσματα θα κριθεί τελικά η αλλαγή του πολιτικού τοπίου. Συνεπώς αναμένουμε τις εκλογές αυτές και θα δούμε ανάλογα με τα αποτελέσματα τι θα γίνει. Εννοείται ότι θα υπάρξουν εκλογικές συμμαχίες. Μετά όμως όλα μπορεί να αλλάξουν, να υπάρξουν δηλαδή διαφορετικές συμμαχίες μετά τη διεξαγωγή των εκλογών. Όσον αφορά τώρα συμφωνία για τις εξαγωγές πετρελαίου, σας είπα ότι ο Πρωθυπουργό μας πήγε στην Βαγδάτη, ότι υπάρχουν συνομιλίες ανάμεσα στον Μπίλ και τη Βαγδάτη για να οδηγηθούμε σε μια λύση που ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Εμείς πηγαίνουμε στις διαπραγματεύσεις αυτές με ελαστικότητα, ευελιξία, αλλά δεν παρετούμαστε από τα συνταγματικά μας δικαιώματα να μοιραζόμαστε και εμείς τους πετρελικούς πόρους της χώρας. Έρχομαι... Για τους χριστιανούς τώρα, αδερφούς μας, στο Κουρδιστάν. Ήταν 10.000 οικογένειες, όπως σας είπα, στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Τώρα πρέπει να είναι 26.000 οι χριστιανικές οικογένειες. Είμαι εναντίον του να φύγουν οι χριστιανοί από το Ιράκ για να πάνε στη Δύση οι χριστιανοί του Ιράκ είναι αυτόχθονες Ιρακίνοι. Τους ανήκει και σε αυτούς η χώρα. Στο Κουρδιστάν έχουμε δώσει όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν σε ειρήνη. Έχουν απόλυτη ελευθερία. Μπορείτε να κάνετε και μια αποστολή εξεταστική για να δείτε ποια είναι η κατάσταση έρευνας, για να δείτε ποια είναι η κατάσταση προσωπικά, αν θέλετε. ο, η κυβέρνηση του Κουρδιστάν δίνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία στους και τα μέσα στους ε, χριστιανούς για να μπορέσουν να μείνουν στην περιοχή μας, ελπίζοντας ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί στο υπόλοιπο τμήμα του, της επικράτειας του Ιράκ. Αν θέλουν να παραμείνουν βέβαια στην περιοχή μας, είναι πάντα καλόδεκτοι. Τους ζητούμε να μην φύγουν όμως από το Ιράκ να μην ξενιτευτούν, να μην μεταναστεύσουν στη Δύση και θα ήταν χρήσιμο και εσείς να τους ενθαρρύνετε να παραμείνουν στο Ιράκ. Ελπίζω λοιπόν ότι έχω δώσει απάντηση σε όλα τα ερωτήματά σας. Ίσως ξέχασα κάτι. Σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε αν ξέχασα κάτι και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ πρόεδρε Μπαζάνη. Και όπως είπα το μήνυμά σας ήταν απόλυτα σαφές. Σε εμά σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο εγχείρημά σας. Στην περιοχή σας και στη χώρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε και έγκαιρος λέει ο πρόεδρος Συνάδελφοι, να προχωρήσουμε. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν κόσμο πολιτισμικών και θρησκευτικών διαφορών. Η συγγήτρια, η συνάδελφός μας, κυρία Μαριά ε, Γιαννάκου, η οποία είναι εδώ και η οποία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η έκθεση αυτή ε, είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας και ανταποκρίνεται πλήρως νομίζω ε, ως ιδέα στα όσα παρακολουθούμε να συμβαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες με την επίδραση των πολιτιστικών και θρησκευτικών διαφορών σε θέματα που αφορούν στις συνεννοήσεις μεταξύ των κρατών μελών με την όξυνση η οποία υπάρχει ε, σε διάφορα ζητήματα, σε πολλές σχέσεις μεταξύ κρατών που άλλοτε διατηρούσαν φιλικές ε, σχέσεις και επικοινωνίες και κυρίως βέβαια με τη χρήση των πολιτιστικών και θρησκευτικών διαφορών και την εκμετάλλευσή της ε, για την ε, όξυνση της επιθετικότητας διαφόρων πλευρών. Βεβαίως η εξωτερική πολιτική της Ένωσης παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και παρά τις προσπάθειες και της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και της Βαρόνης Άστον ε, δεν έχει καταφέρει να είναι ακόμα μια πραγματικά ενιαία πολιτική ακόμη και σε ζητήματα που ε, υποτίθεται ότι συμμερίζονται τις ίδιες αρχές και αξίες ε, τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, προσπάθησα να συνδυάσω στην υπόθεση αυτή τις αρχές τις οποίες βασίζεται η εξωτερική πολιτική της Ένωσης, τουλάχιστον θεωρητικά, γιατί η πρακτική διαφέρει πάρα πολλές φορές, με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας και στα διάφορα πολυμερή φόρα βέβαια. Και όλα αυτά πώς αποδίδουν με βάση την αξιοπιστία, τη συνοχή και τη συνέπεια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς προσλαμβάνονται από τις τρίτες χώρες Επίσης κύριε Πρόεδρε υπάρχει ένα κλίμα το οποίο θα συμπεριλάβω μέσω τροπολογιών στην έκθεσή μου γιατί το μήκος της έκθεσης ήταν περιοριστικό από πλευράς κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που αφορά κυρίως ε, στο διάλογο με τις τρίτες χώρες σε διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό επίπεδο την κατάρτιση του προσωπικού της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για θέματα διαπολιτισμικά και για θρησκευτικό, και διαπολιτισμικό διάλογο, τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σε διάφορα προγράμματα, παραδείγματο χάρη στο πρόγραμμα Αναλίντ, το πρόγραμμα που κάνει το Αναλίντ Foundation ε, και άλλες πρωτοβουλίες ε, διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού χαρακτήρα, όπως το ΚΑΙΣΥΔ στη Βιέννη, με έμφαση στην εκπαίδευση και τη θρησκεία την αξιοποίηση των αντιπροσωπιών της Ένωσης σε όλο τον κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση και την αξιοποίηση των social media. Ε, κύριε Πρόεδρε, πριν από αρκετά χρόνια ε, ο τον ανέπτυξε στο βιβλίο του The Class of the Civilization ε, απόψεις που καλό είναι η δράση μας σημερινή να τις αφήσει έξω από την παρούσα κατάσταση και το παρόν σύστημα. Πριν από 30 χρόνια δεν γνωρίζαμε καν, υποθέτω ότι όλοι μας φοιτώντας στο σχολείο δεν γνώριζαν καν λεπτομέρειες για το ποιες είναι οι θρησκείες που επικρατούν στις αφρικανικές χώρες. Εγώ δηλαδή πρέπει να σας ομολογήσω ότι δεν φανταζόμουν ότι το Ισλάμ έχει τέτοια ευρεία επίδραση στις αφρικανικές χώρες. Σήμερα βλέπουμε να χρησιμοποιείται εξοχήν ο πολιτισμός και η θρησκεία με την εξή θεωρία ότι δήθεν ο πολιτισμός δεν αλλάζει είναι ένα δόγμα, ένα πακέτο που δεν αλλάζει, ενώ όλοι ξέρουμε ότι αλλάζει, εξελίσσεται ο πολιτισμός. Και η θρησκεία δεν αλλάζει και επομένως ζητήματα που φέρονται ως δογματικά και που έχουν ρυθμιστεί ε, στα βάθη των αιώνων δεν μπορούν να αλλάξουν. Άρα αφού δεν μπορούν να αλλάξουν δεν μπορεί να υπάρξει ανεκτικότητα, δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση και δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη στο πλησίασμα των διαφόρων πλευρών. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα πολύ αρνητικό για τους λαούς των οποίων οι ηγεσίε συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Θα σας έλεγα είναι εγκληματικό και χαρακτηριστικά αυτό φαίνεται στη μεταχείριση των γυναικών τον οποίον το στάτους δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη οντότητα σε πολλές από τις χώρες αυτές ή τις κοινότητες ή τις κοινωνίες δηλαδή μέσα σε χώρες που τυπικά είναι δημοκρατικές από πλευρά νομοθετικής υπάρχουν κοινότητες που αγνοούν και παραμερίζουν κάθε σύστημα νομικό που εξασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ότι η δημιουργία σταθερών δημοκρατιών που προσφέρουν ελευθερία στους πολίτες τους είναι το καλύτερο όπλο για την οικοδόμηση της ειρήνης και φυσικά για τη συνεργασία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και προς το συμφέρον σε τελευταία ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Άρα ο δημοκρατισμός των διαφόρων χωρών είναι σημαντική ε, βασική αρχή και βλέπουμε ότι πιο πρόσφατα σε εξεγέρσεις όπως την Αραβική Άνοιξη ε, η εξέγερση αφορούσε και την αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη οντότητα και τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. Άρα δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μόνο στη Δύση ή μόνο στην Ευρώπη οι λαοί είναι φτιαγμένοι για τη δημοκρατία. Γιατί ακούγονται και αυτές οι απόψεις. Ότι δηλαδή είναι τέτοια η κατάσταση ε, πολιτισμικά και θρησκευτικά σε ορισμένες χώρες ώστε οι λαοί αυτοί δεν μπορούν να κυβερνηθούν εν δημοκρατία. Αντίθετα, διάφορες εξεγέρσεις δείχνουν το αντίθετο. Και βέβαια αυτό οφείλεται στην κοινωνία της πληροφορίας και τις γνώσεις κύριε Πρόεδρε που είναι και η μεγαλύτερη επανάσταση κατά τη γνώμη μου ε, της εποχής μας γιατί δίνει ευκαιρίες σε ανθρώπους και σε λαούς και σε ε, οντότητες που δεν θα μπορούσαν ούτε θα γνώριζαν τι γίνεται πέρα από το χωριό τους ούτε θα μπορούσαν να επικοινωνούν και θα ήταν βέβαια κάτω από την μάστιγα αυτών των αντιλήψεων που περιέγραψα πριν ενώ τώρα μπορούν κάλλιστα να επικοινωνούν με όλο τον κόσμο. Επομένως προσφέρονται τα social media, το ίντερνετ και η κοινωνία της πληροφορίας. Ασχέτως εάν προσφέρονται και για το κακό. Προσφέρονται όμως και γι' αυτό. Τώρα, η προάσπιση πολιτισμών μικροτέρων κοινοτήτων και μειονοτικών πολιτισμών και η ενίσχυση ε, του δικαιώματός τους να εκφράζονται ελεύθερα είναι επίσης ένας τρόπος για να μην αντιμετωπίζονται οι πολιτισμικές διαφορές ως αντιπαράθεση ασυμφιλίωτων συνασπισμών. Επομένως, καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την κύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτισμικών εκφάσεων και τονίζει τη σπουδαιότητα που έχει η πολιτισμική διπλωματία και η πολιτισμική συνεργασία. Παρατηρούμε ότι η κλασική εξωτερική πολιτική όπως τη γνωρίζαμε πριν από πολλά χρόνια ε, έχει μεταβληθεί. Φυσικά είναι τα οικονομικά συμφέροντα αλλά είναι και άλλες διαδικασίες και άλλοι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και να κάνουν ουσιαστικότερες τις σχέσεις μεταξύ λαών με διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετική θρησκεία. Στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ιδίω στο ε, Συμβούλιο Ασφαλείας, ε, δεν αντικατοπτρίζονται με τον κατάλληλο τρόπο, δεν αντικατοπτρίζεται η πολυμορφία των παγκοσμίων παραγόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια και τα κράτη-μέλη τελούν εν συνεννοήσει και βρίσκουν έδαφος για διάλογο και συνεργασία με τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών ώστε να βρεθούν λύσεις που είναι πάνω από πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές. Αλλά οι εντάσεις και τα αδιέξοδα που παρεμποδίζουν την εξέβρεση αυτών των λύσεων προκύπτουν από την αντίδραση κρατών σε συμφωνίες αυτού του είδους. Κυρίως λόγω στρατηγικών συμφερόντων και όχι λόγω αντικρουωμένων ηθικών αξιών. Επίσης η θεωρία που επικρατεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και στα στρατηγία της εξωτερικής πολιτικής, σε πολλές από τις χώρες μας είναι, τι να κάνουμε, αυτές είναι παραδόσεις, είναι πολιτισμικές διαφορές, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή πολλές φορές ισχυριζόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για το ότι οι γυναίκες στην κυριολεξία δολοφονούνται στις χώρες της Αφρικής και γιατί τελούν σε μια κατάσταση που είναι χειρότερη ακόμα και από την κατάσταση των ζώων. Και όμως μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να το κάνει διότι εδώ έχουμε προκλήσεις θρησκευτική επιρροής στη διεθνή πολιτική σκηνή συνεχώς. Δηλαδή πέρα από τους κινδύνους που δημιουργούνται από την τρομοκρατία η μεγαλύτερη κίνδυνη είναι η διάδοση των ιδεών, της οξύτητας, της συνεχούς αντιπαράθεσης, της έλλειψης ανεκτικότητας, συνδυασμένες δήθεν με θρησκευτικέ οδηγίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί φυσικά με τα Ισλαμικά κράτη και καλό είναι να ξεκινήσει από τα κράτη που δεν έχουν τόσο υπερβολική φονταμεταλιστική προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων και έχουν μια αντίληψη του Ισλάμ που δεν είναι με τόσους αποκλεισμούς. Για να υπάρξει μια παρεμπόδιση της προώθησης των θρησκευτικών ερμηνεών σε όλα τα φαινόμενα της φύσης, την επιστήμη παντού, να δίνονται θρησκευτικές ερμηνείες. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, για να έχουμε αξιοπιστία, συνοχή και συνέπεια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουμε και υποδειγματική στάση της Ευρώπης. Πρέπει να καταργηθούν όλα τα νομοθετήματα που αντιβαίνουν σε όσα αναφέρθηκαν πριν. Πρέπει να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να προωθήσει την ελεύθερη έκφραση, την ελευθερία του τύπου και την ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένοι εκπρόσωποι της να θεωρούν τις ε, πολιτικές εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως δήθεν παραδόσεις που προέρχονται από τα βάθη των αιώνων, από τη θρησκεία κλπ. Πρέπει να δώσουμε μάχη, επομένως, ε, για αυτά που πιστεύουμε και για ένα πιο ελεύθερο κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. κυρία Λιούψεβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα βουλγάρικα θα απευθυνθώ στην εισηγήτρια. Η έκθεση αυτή προσπαθεί να ανατάμει τις κύριες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση πολιτιστικών και θρησκευτικών διαφορών και επικοινομορφιών. Αυτά τα οποία παρουσίασε η κυρία Γιαννάκου μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια σωστή προσέγγιση για το θέμα αυτό η έκθεση αντιμετωπίζει τα κύρια έγγραφα τα οποία καθορίζουν τη στάση που πρέπει να ισχύει έναντι της διαφοράς και των διαφορετικών πολιτισμικών πραγματικότητων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς θα τίθενται σε εφαρμογή όλα αυτά τα έγγραφα, ώστε να μπορέσουν με τον τρόπο αυτό να προστατεύσουν όλες τις ανθρώπινες αξίες. Στην έκθεση όμως δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε για μια νέα διεθνή τάξη. Απλώς θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην, ε, στο κράτος δικαίου, στην προστασία των μειονοτικών ομάδων και στην ανεκτικότητα εναντί τους. Αυτά είναι και η βάση μιας μεγαλύτερης συνεργασίας <clears throat> μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, τις διακρίσεις και όλα αυτά τα αντιπαραγωγικά στοιχεία που προκύπτουν από τις ε, διακρίσεις και που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προφανές βέβαια ότι υπάρχουν διαφορετικά πολιτισμικά θεμέλια για τους πληθυσμούς και τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια δημοκρατική αντιμετώπιση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια θετική αντιμετώπιση σε σχέση με τρίτους λαούς και τρίτες χώρες όταν είναι διαφορετικοί από μας. Δυστυχώς υπάρχουν ποικίλε συμπεριφορές στην Ευρώπη έναντι άλλων θρησκειών. Αυτό δεν είναι συμβατό με αυτά τα οποία έχουμε δεχτεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να γίνουν δεκτές αυτές οι αξίες και θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ακεραιόφρονες στάσεις οι οποίες δεν δέχονται τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως δεν μπορούν να γίνουν δεκτές και από εμά. Θα να δω να αναφέρονται και περισσότερο στην έκθεση για την επιρροή της θρησκείας σε πολιτικές διαδικασίες λήψης απόφασης και έχουμε προκλήσεις στον τομέα αυτό στις εξωτερικές πολιτικές μας. Θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες όμως σε αυτές τις διαδικασίες για να είμαστε πιο επιτυχείς. Βλέπουμε και σε άλλα μέρη του κόσμου ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα προσπαθήσει, δεν θα πρέπει να προσπαθεί να εξάγει τις δικές της αξίες, αλλά αντίθετα να δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο για να μπορέσει να πριτανεύσει η ανεκτικότητα και οι καλές σχέσεις με τους εταίρους μας και με όλες τις τρίτες χώρες. Πιστεύουμε ότι με τις τροπολογίες που θέτουμε θα συμβάλλουμε περαιτέρω στην ποιότητα της έκθεσης, ώστε να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και να μπορεί έτσι να προασπίζεται τις αξίες μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νικολάτη. Ευχαριστώ, κυρία Νικολάτη, ευχαριστούμε. Ε, θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή αφορά και την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό κόσμο. Μας ενδιαφέρει το ευαίσθητο λοιπόν αυτό θέμα, γιατί χρειαζόμαστε μια ισορροπή προσέγγιση. Ιδάλλως, ε, διακινδυνεύουμε να θεωρηθεί ότι ε, κοιτάζουμε με μεροψία τον υπόλοιπο κόσμο και έτσι εξετάζουμε τι πολιτιστικέ και θρησκευτικέ διαφορέ. Πιστεύω λοιπόν ότι στην έκθεση αυτή πρέπει να αποφύγουμε την τροπολογία ε, περί ριζοσπαστικοποίηση δεν θα πρέπει εμείς να λάβουμε θέση κατά του φονταμενταλισμού. Δεν είναι αυτός ο λόγος ύπαρξης της έκθεσης, αλλά προκειμένου να προωθήσει την ανεκτικότητα και την ανοχή, ε, μια από τις πρωταρχικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η ανεκτικότητα να διαδοθεί και στον υπόλοιπο κόσμο. Διότι ακριβώς πρέπει να αποδεχτούμε ότι πολυμορφία στον κόσμο σημαίνει διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές νοτροπίες. Νομίζω ότι δεν είναι η στιγμή να εντοπίσουμε συγκεκριμένα θρησκευτικέ ομάδες ως απειλές. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για το φουνταμενταλισμό και πιστεύω ότι στόχος της έκθεσης αυτής θα πρέπει να είναι να αποδείξει ότι ο πρωταρχικός στόχος της εξωτερικής μας πολιτικής είναι η ανεκτικότητα να προωθηθεί μέσω της διεθνούς συνεργασίας από νομική σκοπιά τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε πολλά στοιχεία στο πλαίσιο της σύμβασης του ΙΕ, διότι μιλήσαμε για τις σχέσεις με τρίτες χώρες, αλλά πολλές από τις χώρες αυτές είναι συμβαλόμενα μέρη της Γενικής Σύμβασης του ΙΕ. Πολλοί έχουν προσπογράψει και τις ειδικότερε συμβάσεις για τα δικαιώματα των πολιτών και το καθεξής. Αυτό το κεφάλαιο πρέπει να είναι ένα κεφάλαιο όπου θα υπάρξει βελτίωση για το λόγο αυτόν θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια ανοιχτόμυαλη, ανεκτική, διαλλακτική στάση στα πράγματα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Έπειτα θα έχουμε αρκετές τροπολογίες να υποβάλλουμε, όμως καλώ τους συναδέλφους στην έκθεση αυτή να τηρήσουν πραγματικά ισόρροπη στάση. Διότι μπορούμε να θίξουμε πολλαπλά ζητήματα για το κατά πόσον είμαστε ανώτεροι ή όχι, αλλά η έκθεση αυτή δεν έχει αυτό στόχο. Έχει να κάνει με την αξιοπιστία μας. Σας ευχαριστούμε κύριος Πέτερλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η συνάδελφος ε, κυρία Γιαννάκου αποφάσισε να συντάξει έκθεση για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Θέμα το οποίο ε, δει όλες τις απαραίτητες προσοχής μας. Ε, εδώ έχω δει από προσωπική μου πείρα πόσο ευαίσθητο μπορεί να είναι ένα τέτοιο θέμα και πραγματικά έχουμε ζήσει από κοντά το πόσο ευπρόσδεκτη είναι ανοιχτό μια λιστάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τις θρησκευτικέ διαφορές λόγου χάρη. Είχαμε επανειλημμένως ε, συναντήσεις με πολλές ομάδες στην Επιτροπή μας και δεν θεωρούμε ε, ότι η βία είναι ένας τρόπος να λύνονται διαφορές λόγου χάρη. Τώρα μιλάμε για ανεξιθρησκεία, για διώξεις των χριστιανών εδώ νομίζω αυτά πρέπει να αποτελούν μέρος της φραγίδας της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η θρησκεία να μην είναι κάτι που το εξετάζουμε από ιδεολογική σκοπιά όπως το παρελθόν, αλλά να, να αντιμετωπίζεται ως ομάδα ατόμων με διαφορετική ταυτότητα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κοινωνίας, μιας ευρύτερης κοινότητας. Ως ε, εισηγητής λοιπόν ε, ελπίζω η εισηγήτρια να στηρίξει την ενιαία και συνεκτική πολιτική στα θέματα αυτά στο πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό μας περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτού του διαλόγου μάλιστα δεν θα πρέπει να πάψουμε να αντιδρούμε στα παρουσιαζόμενα προβλήματα, αλλά να μπορούμε να λάβουμε και μέτρα στρατηγικής σημασίας. Και ολοκληρώνοντας να πω ότι θα πρέπει να δοθεί σημασία στα ε, να αποφύγουμε μάλλον τα βιαστικά συμπεράσματα και του χαρακτηρισμού για τι θρησκευτικέ διαφορέ. Αυτοί κάποιε φορέ εξυπηρετούν πολιτικέ σκοπιμότητε απλώ και δεν ε, είναι προ το συμφέρον των πολιτών και σε καμία περίπτωση δεν έχει κανένα νόημα να ονομάζουμε συγκεκριμένε ομάδε του πληθυσμού φονταμενταλιστέ ή τρομοκράτε. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γιαννάκου και πάλι, εάν θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή δεν έχει σκοπό να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία δεσμενής αναφορά σε άλλες θρησκείες. Προφανώς η έκθεση προωθεί το, μιλάει για διαθρησκευτικό διάλογο και για διαπολιτισμικό διάλογο. Όμως δεν μπορούμε να αποκρύψουμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί θρησκείες ε, για άλλους σκοπούς και για άλλους λόγους και ότι εκεί ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές συναντάει ένα τείχος ασυνεννοησίας. Βέβαια μπορεί να μου πείτε ότι ο καθένας έχει τις απόψεις του και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τότε δεν πρέπει η Ένωση να ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ κόλλησε η, έκθεση, η συμφωνία με τον Καναδά επί μήνες, διότι ζητούσαμε τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι εκπρόσωποι του Καναδά έλεγαν ότι ο Καναδάς τα εξασφαλίζει καλύτερα από την Ένωση και δεν δέχεται να τα βάλει μέσα στο κείμενο. Επομένως, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου να αφαιρέσουμε το φονταμενταλιστές. Είναι μια πραγματικότητα. Εάν θέλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχει αυτό, τότε δεν έχει λόγο και η έκθεση. Για ποιο λόγο να υπάρχει η έκθεση αφού όλα πάνε καλά, αφού ε, όλες οι θρησκείες συνεργάζονται μεταξύ τους αφού εξασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή δεν είναι αλήθεια όμως. Αυτό δεν είναι αλήθεια καθόλου κύριε Πρόεδρε. Και εγώ δεν σκοπεύω να κάνω μια έκθεση ψεύτικη. Θυμάμαι πολύ καλά στη δεκαετία του 80 κάποτε συμμετέχοντας στο ΑΣΕΠΕ κατέφθασαν αφρικανικής χώρας εκπρόσωποι όπου ήταν τρεις γυναίκες υπουργοί και ένας άνδρας τις γυναίκες τις είχαν ορίσει τρεις μέρες πριν και τις ξύλωσαν τρεις μέρες μετά. Και ήρθαν σε αυτές τις αίθουσε για να μας πούν ότι είναι πιο δημοκρατικοί από τους Ευρωπαίους γιατί έχουν ορίσει τρεις γυναίκες υπουργού. Λοιπόν, να μην, ε, ε, ε, τα τελευταία χρόνια οι θρησκείες έχουν χρησιμοποιηθεί ως μοχλή καταπίεσης και βασανισμού και ιδιαίτερα των γυναικών. Και αυτό δεν μπορεί να το αποκρύψει η έκθεση. Εάν όλα πάνε καλά τότε τι νόημα έχει η έκθεση. Λοιπόν ας κάνουν τις τροπολογίες τους όλοι, όποιες θέλουν. Εγώ θέλω να σας πω το χρονοδιάγραμμα που είναι 10 Φεβρουαρίου θα συζητήσουμε για δεύτερη φορά. Στις 11 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Και βέβαια μέχρι τις 23 δηλαδή μεθαύριο υπάρχει περιθώριο να γίνουν τροπολογίες θα τις συζητήσουμε όλοι μαζί θα τις συζητήσουμε με τους σκιώδεις συζητητές για να υπάρχει μια έκθεση η οποία δεν θα ειδωθεί αρνητικά δηλαδή στην έκθεση δεν αναγράφεται πουθενά ότι έχουμε καμία εναντίωση σε κάποιες θρησκείες όλες οι θρησκείες είναι σεβαστές αλλά κύριε Πρόεδρε εάν υπό το πρόσχημα μιας θρησκείας πολιτικές ηγεσίε και εξουσίες α, λειτουργούν ολοκληρωτικά και δικτατορικά δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε αυτό ή να διαφορήσουμε. Σας ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 23 Ιανουαρίου στις 12 η ώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Έχουμε κλείσει την ε, τακτική συνεδρία. Περνάμε τώρα στην και κλεισμένων των θυρών. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα να είναι παρόντες στην ε, συνεδρία και κλεισμένων των θυρών, τους εξωτερικούς παρόντες να αποχωρήσουμε και να συνεχίσουμε και κλεισμένων των θυρών.